Επομένως, ε, θα συζητήσουμε με τους ε, συντονιστές ε, τι θα κάνουμε στο μέλλον με την πρόταση ψηφίσματος που έχουμε μπροστά μας όσον αφορά το transmission charging. Ας συζητήσουμε καταρχάς πώς θα έχει διαδικασία σχετικά με την ψηφοφορία. Ο κύριος Ρούμπικ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σουάποντα όμω είναι στην αίθουσα, στο βάθος της αίθουσας. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ακούστε πολύ προσεκτικά πώς έχει το ζήτημα αυτό πρέπει να δούμε αν θα ψηφίσουμε αυτή την πρόταση ψηφίσματος ή όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Κύριε Σουόμπο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ρούμπικ ε, φτάνει αυτή τη στιγμή από το αεροδρόμιο. Το ζήτημα όντως είναι πολύ λεπτό μια ένσταση σε σχέση με τη διαδικασία επιτροπολογίας, ακόμα και αν δεν έχουμε την επιτροπολογία επίσημα, για οικονομικούς λόγους. Η άποψη που έχουν κάποιοι από εμά και ξέρω φυσικά ότι είναι διάφοροι που την έχουν, δεν είναι θέμα κομματικών, ε, κομματικής τοποθέτησης. Όμως σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δίκιο αφενός νομικά δεν έχει δίκιο και δεν έχει επί της ουσίας δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση περί τίνος πρόκειται για το ότι θα πρέπει να ε, αποζημιωθούν σε σχέση με τους μετασχηματιστές ε, για τη διαβίβαση ηλεκτρικής ενέργειας. Για εκείνες τις χώρες ε, που περνά το ηλεκτρικό ρεύμα από εκείνες. Αν σκεφτούμε ότι οι DSOs έχουν, πρέπει, έπρεπε να κάνουν μια σειρά επενδύσεων και αυτό είναι αποφασιστική σημασία για το μέλλον, για το δυναμικό δηλαδή του δικτύου που θα πρέπει να αναπτυχθεί, εμείς πιστεύουμε ότι τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται στο Ταμείο δεν επαρκούν. Δεύτερον, είναι και κάπως προβληματικό ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάποιους πολύ γενικόλογους, αφηρημένους ε, γενικόλογους λόγους ε, ως επιχείρημα βασίζεται σε αυτούς και ότι κατά τα τέλη του 2010, τα τέλη αυτού του έτους θα δώσει εντολή να συνταχθεί μια μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξεταστεί τι συμβαίνει με τα δεδομένα δικαιολογημένα κόστη μεταφοράς. Δεν θέλω να πω ότι είναι το αποφασιστικό επιχείρημα ότι το ποσό είναι υπερβολικά χαμηλό, αλλά τα βάθρα, η βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λυπή, έχουν ατέλειες και σε περίπτωση που τίθεται η έγκριση αυτού του ψηφίσματος σήμερα, ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γοργά να καταλήξει σε άλλη βάση λήψης απόφασης και να έχουμε μια βιώσιμη αντιληπτή με βάση κάποια νομική βάση που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή για το κόστος και την αντιστάθμιση και αποζημίωση όσον αφορά τα, ε, τα DSO. Αυτό είναι το αποφασιστικό νομίζω επιχείρημα και όχι το επιχείρημα το ποσό είναι μικρό. Σας ευχαριστώ. Εσείς συνάδελφοι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το θέμα, αν ψηφίσουμε το ψήφισμα, εγώ ζητώ Πέντε λεπτά όλα και όλα για να μπορέσω να μιλήσω με τα μέλη της ομάδας μου. Γιατί η ομάδα μου δεν μπόρεσε να συζητήσει αυτό το θέμα, Πρόεδρε. Και γι' αυτό αυτό συνέβη. Δεν το έχουμε συζητήσει. Χρειαζόμαστε, ζητάμε πέντε λεπτά τουλάχιστον. Μου λένε υπάρχουν ομάδες που έχουν αποφασίσει free vote, ελεύθερη ψήφο. Εγώ συντονίστρια δεν μπορώ να πάρω μια τέτοια απόφαση για την ομάδα μου όμως, γιατί δεν είχαμε ούτε την ελάχιστη ανταλλαγή απόψεων. Λοιπόν, ή δεν θα ψηφίσουμε ή αν θα ψηφίσουμε χρειαζόμαστε και είναι αυτονόητο αυτό κάποιο χρόνο για να συζητήσουμε και σχολιάσουμε τα θέματα. Σε ευχαριστώ. Η διαδικασία δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο επειδή η αντίρρηση του κυρίου Ρούμπιχ, συναδέλφου και του κυρίου Σβόμποντα υπήρχαν και την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τους συντονιστές ενημερωθήκαν, ε, έδωσαν ειδοποίηση ότι σε σχέση με τη γραμματεία θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για ένα ψήφισμα. Αν θέλουμε να πούμε κάτι και αν θέλουμε να τονίσουμε κάτι, σήμερα πρέπει να το κάνουμε ώστε να περάσει στην Ολομέλεια έγκαιρα. Αλλιώς δεν θα είναι δυνατόν. Είναι το θέμα τη ίδια τη διαδικασία που απαιτεί αυτό. Αλλά νομίζω θα βρούμε μια βιώσιμη λύση. Το επόμενο ο κύριο Τούρμες, παρακαλώ. Ε, Βρίσκω αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εμεί τα θέματα και που ο συνάδελφο Βόμποντα έθιξε, θα έπρεπε να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει σε αυτό και να μας πει την άποψή της, να μας εξηγήσει κάπως για εκείνους που δεν έχουν εξοικειωθεί σε βάθος με το θέμα τι συμβαίνει και περί τίνος πρόκειται να μας πει. Πρόεδρος, έχω τρεις που έχουν ζητήσει τον λόγο. Ερώτηση, να δώσουμε πρώτα τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι λέτε. Γιατί θα μπορούσε να είναι ευφυές σε σχέση με σας ε, κυρία Έκα ε, Μαντουρέλ, κύριε Τσίτσεστερ, να πάρει τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε θα διευκολυνθούν τα πράγματα. Αν συμφωνείτε και δεν έχετε αντίρρηση. Ο κύριος Ομπράιν λοιπόν έχει τον λόγο από την Επιτροπή για μια σύντομη αποσαφήνιση των πραγμάτων. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Uh, thank ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι αυτή, ε, αυτό το θέμα των αντισταθμίσεων είναι κάτι που το, το έχουμε, μας έχει απασχολήσει από την αρχή της συζήτηση για το θέμα αυτό. Ήδη από το 97 νομίζω έχει ξεκινήσει να συζητιέται. Οπότε δεν έχουμε καταλήξει σε δικά μας συμπεράσματα. Αυτό το σύστημα αντισταθμίσεων, intertransmission, σκοπό έχει να επιφέρει ισορροπία στην εσωτερική αγορά και να επιτρέψει ένα σύστημα μετάβασης στην Ευρώπη. Το 2003 με τον κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια υπήρχε μια διάταξη για αποτελεσματικούς ως προς το κόστος, διαφανείς και σταθερούς κανόνες που προβλέπονταν αντισταθμίσεις αυτού του τύπου και προβλεπόταν η εισαγωγή τους με τη διαδικασία τη επιτροπολογία από την Επιτροπή. Όμως επί 7 χρόνια αυτό ίσχυε σε οικειοθελή βάση μεταξύ των συστημάτων που ήθελε να συνεργαστούν. Και δεν γίνονταν συνεχώς Ναι, και γίνονται μάλλον συνεχώ συμφωνίε, οπότε η Κομισιόν υιοθέτησε κατευθυντήρε γραμμέ το 2007. Το 2008, 2007 μάλλον και 2008 η Επιτροπή εξέτασε το θέμα αυτό. Ολοκλήρωσε ένα γύρο δημοσίων διαβουλεύσεων. Ολοκλήρωσε κατά τη διαδικασία διαβούλευση με του ε, ενδιαφερομένου στο φόρουμ τη Φιλανδία, όπω ονομάστηκε το 2009 και υπέβαλε τις προτάσεις της μέσω της Επιτροπολογίας, ατύπως πέρσι τον Δεκέμβριο και επισήμως φέτος τον Μάρτιο. Υπήρξαν δύο διδικασίες επιτροπολογίες που είχαν σχέση με το θέμα αυτό. Μία μας απασχολεί όμως σήμερα. Αλλά σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι όλα αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν από την 3η Μαρτίου 2011, όταν ο κανονισμός 2028 εκπνέει, εκπνέψει μάλλον, και ελπίζουμε ότι θα αντικατασταθεί από ένα νέο κανονισμό της Επιτροπής και ένα νέο νομοθετικό πακέτο ενδεχομένως. Θα πρέπει ίσως να δούμε τους δύο κανονισμούς της Επιτροπής από κοινού και σημαντικό είναι ο ρόλος του οργανισμού να αποτιμήσει το κόστος και να δει τι γίνεται με την χρήση των συστημάτων αυτών διασυνοριακά. Και βεβαίω το ίδιο κόστο πρέπει να αποτιμήσουν και οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ, ώστε να διαθέσουν τι υποδομέ αυτέ εντό των κρατών μελών. Μέχρι ο οργανισμό να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά και να μπορεί να φέρει πέρα το έργο αυτό, έχουμε προβλέψει ένα κόστο για τη διάθεση των υποδομών 100 εκατομμυρίων Και αυτό αφού συζητήσαμε με τους εμπειρογνώμονες και τους υπευθύνους των συστημάτων μετάδοσης ενέργειας Και βεβαίω εκπροσωπήθηκαν στι συναντήσει αυτέ τόσο τα κράτη-μέλη όσο και η Επιτροπή. Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή θα είναι πολύ σημαντική και θα μα επιτρέψει να δώσουμε έναν επιτυχημένο επίλογο σε μια ιστορία που έχει τραβήξει πάρα πολύ καιρό τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Η κυρία Έκα έχει τον λόγο, η συνάδελφος στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα το κείμενο του ψηφίσματος θα έπρεπε να διανέμηθει ένα αντίτυπο στα μέλη για να μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα όπως η κυρία Πιλάντερ Καστίγιο προτείνε και θα υποστηρίξω το ψήφισμα εφόσον ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Also, Πρόεδρος. Θα κάνουμε και κάποια άλλα πρόσθετα αντίγραφα και θα δοθούν στα μέλη. Είχαν ήδη αποσταλεί χθε. Η κυρία Μαντουρέλ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μια απόφαση. Κάναμε τις αντίστοιχες διαβουλεύσεις που έπρεπε και πράγματι η δική μα λοιπόν θα ήταν ελεύθερης ψήφου μια και υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να υπάρχουν κάποιοι να τοποθετηθούν εναντίον. Αλλά στο επίπεδο των κρατών μελών είμαστε διαιρεμένοι ούτω ή άλλω. Εν πάση περιπτώσει, θα σα έλεγα ότι η κυρία Καστίγιο έχει δίκιο. Εντάξει, στου συντονιστέ σα αποφασίστηκε να γίνει συζήτηση για ένα σχέδιο που έπρεπε να προετοιμάσει η Γραμματεία. Όμω ε, δεν έγινε λόγο για ψηφοφορία για οποιαδήποτε στιγμή. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθούν αυτά τα θέματα και να οριμάσουν. Απ' την άλλη πλευρά κατανοώ ότι είναι αναγκαία να ληφθεί μια απόφαση το δυνατόν νωρίτερα για αυτό το θέμα. Και έτσι υπάρχει αυτή η πίεση που έθεσε ο Πρόεδρος να τοποθετηθούμε. Εγώ το είπα ώστε να αρχίσει στην ομάδα μας μετά από διαβούλευση με τις ε, νομικές υπηρεσίες και του τους ε, ε, πραγματογνώμονες δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε αντίθετοι. Εκείνο όμως το οποίο συμβαίνει είναι ότι είναι οι ίδιες οι ρυθμιστές, οι ίδιες οι υπηρεσίες αυτές είναι διαιρεμένε, είναι διχασμένες και αυτό για διαφορετικού λόγους. Για μας είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι guidelines, οι κατευθυντήρες γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι προσωρινού χαρακτήρα. προβλεπετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει μια μελέτη ή θα κάνει μια αξιολόγηση πιο ρεαλιστική για το κόστο όσον αφορά τα τέλη του 2010. Και εμεί θα θέλαμε να αναμείνουμε να δούμε αυτή την ε, τελική αξιολόγηση. Αυτή είναι η θέση μα Πρόεδρε. Καταρχήν η ομάδα μα ε, είναι υπέρ τη free vote, ελεύθερη ψήφου. Λαμβάνοντα όμω υπόψη αυτά τα στοιχεία τα οποία σα ανέφερα. Ευχαριστώ. Ε, Κύριος παρακαλώ. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να βιαστούμε και να το μετανιώσουμε στη συνέχεια. Επομένως, προτείνω να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία όπως προβλέπεται στη μερίσια διάταξη, πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε το χρόνο μετά όσοι επιθυμούμε να κάνουμε διαβούλευση, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επομένω, συμφωνώ με την κυρία Καστήλοβέρα ότι θα πρέπει να γίνει μια σύντομη διακοπή προκειμένου να μας δοθεί δυνατότητα να συνεδριάσουμε με τις πολιτικές ομάδες και στη συνέχεια να ξανασυνεδριάσουμε και να ψηφίσουμε την πρόταση. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να μας δοθεί λίγος χρόνος προκειμένου να διεξαχθεί μια συζήτηση και κατά αυτόν τον τρόπο θα είμαστε και πιο ικανοποιημένοι με την ψηφοφορία, πιστεύω. Μπορεί να γίνει αυτό αργότερα στη σημερινή συνεδρία, αργότερα σήμερα. Ο κύριο Βιντερ Κουαντάς. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα θέμα από αυτά που είναι χαρακτηριστικά δύσκολο να βρεθούν θέσει ομοιογενείς μέσα στου κόλπου των ομάδων. Επειδή έχουμε μια κατάσταση εδώ που έχει οδηγεί σε σύγκρουση θεμητών συμφερόντων μεταξύ χωρών που θα λέγαμε διαμετακόμισης και χωρών που δεν είναι χώρες διαμετακόμισης, αλλά είναι χώρες ή υποδοχής ή αποστολής. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά είπε η κυρία Καστίγιο πιο πριν, η ομάδα του ΕΛΚ βρίσκεται σε μια παρόμοια κατάσταση όπως οι άλλες ομάδες, όπως στους κόλπους της ομάδας του ΕΛΚ υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Και γι' αυτό δεν μπορούμε τώρα να τοποθετηθούμε χωρίς πιο πριν να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω πρόεδρε είναι το εξής. Είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να, να έχει κανείς αντιρρήσει σε σχέση με τη διαδικασία για την επιτροπολογία υπό όρους ε, διαδικασίας. Γιατί η νομική μας υπηρεσία ήταν αρκετά σαφής ότι ήταν σωστή η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί δεν εξαντλείται όμως η πολιτική στις διεργασίες και στις διαδικασίες, Πρόεδρε. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία ακολουθούν. Όμως, μια τέτοια επικέντρωση στη διαδικασία δεν έχει μεγάλο μέλλον και προοπτικές. Τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να αξιολογηθούν, χωρίς αμφιβολία. Και αυτό πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε. Εντάξει, όμως, εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε, όσον αφορά το ΕΛΚ, και το είπε και η συντονίστρια μα χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο χρόνο να προβληματιστούμε από κοινού. Προτού λάβουμε μια θέση και υιοθετήσουμε μια θέση. Mr. Rübich. Κύριος Ρούμπιχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα <clears throat> να ζητήσω συγγνώμη, είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο μου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση, θέμα αρχή, διότι τώρα γνωρίζουμε ότι μέσα από τη συνθήκη τη Λισαβόνα φυσικά η επιτροπολογία αποκτά μια νέα ε, σημασία. Και έτσι εμείς ως Κοινοβούλιο σε Ευρωβουλή είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε, να δούμε αν αυτά που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο πραγματικά ανταποκρίνονται στο ενισχύει δίκαιο και σε αυτή την περίπτωση πιστεύω υπάρχει αντιφάσκη η ε, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, στο θέμα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Χρειαζόμαστε την ενιαία εσωτερική αγορά. Δεν είναι δυνατόν κάτι που διαβιβάζεται, μία διαβίβαση να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με το ό,τι γίνεται σε ένα κράτος μέλος. Αυτό για τις ε, χώρες που βρίσκονται ε, στις άκρες, στις παρυφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα αν η Ολλανδία, η Φινλανδία, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα και για την εξαγωγή αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας. Διότι ζητείται να γίνουν επενδύσεις ε, για να είναι βιώσιμο το δίκτυο και πρέπει να αποσβεστούν αυτές οι επενδύσεις. Δεν είναι δυνατόν ε, να γίνει αυτό χωρίς να υπάρξουν επενδύσεις. Θα υπάρξουν προσκόμματα και εμπόδια. Και αυτή η απόφαση παραβιάζει και αντιβαίνει στις αποφάσεις και την αρχή της ενία εσωτερικής αγοράς. Ο κύριος Τούρμες, παρακαλώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα όπου η Αυστρία παίρνει πολύ συχνά το λόγο, ακριβώ γιατί θα χάσει πολλά χρήματα. Οι Ισπανοί επίση ζητάνε συχνά το λόγο γιατί θα κερδίσουν από αυτή την ιστορία. Η χώρα μου, το Λουξεμβουργό, δεν είναι χώρα μεγάλη διέλευση, ούτε μεγάλο εισαγωγέα, ούτε εξαγωγέα. Δεν έχω λοιπόν κανένα ιδιαίτερο συμφέρον στην όλη υπόθεση, όμω έχω δύο παρατηρήσει. Αυτή ήταν η δική μου εισήγηση. Ε, έχω δύο παρατηρήσεις λοιπόν. Πρώτον, το βρίσκω λίγο παράξενο να το χρειαζόμαστε αυτό τώρα για να αλλάξει ο κανόνας δηλαδή σε μια μεταβατική περίοδο ενώ συστήνουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ρυθμιστών η οποία θα είναι στην, ε, ο καταλληλότερος φορέας για να ορίσει τους σωστούς αριθμούς τις σωστές ποσότητες. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί πρέπει να αλλάξουν ε, οι κανόνες φέτος. Και έπειτα Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σέβεται κάπως περισσότερο το σώμα μας, διότι εάν το θεωρούν τόσο σημαντικό, θα έπρεπε να έχουν προσπαθήσει από λίγο καιρό νωρίτερα να μας εξηγήσουν περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί αυτό ίσω να δώσει και ένα μάθημα, για παιδαγωγικού λόγου, δηλαδή, προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το πώ πρέπει να συμπεριφέρεται. Σα ευχαριστώ πολύ. Και έτσι περιγράψαμε το πρόβλημα. Έχουμε διαδικαστικά ένα πρόβλημα, επειδή πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα, ώστε να καταλήξει στην Ολομέλεια και έχουμε πιεστικές προθεσμίες. Από, από την άλλη πλευρά κατανοώ τους άλλους συναδέλφους που είπαν ότι χρειάζεται χρόνος για να συζητηθεί το θέμα. Εδώ Τώρα δύο δυνατότητες έχουμε. Ή θα ψηφίσουμε τώρα ψηφίζοντας στον χρόνο ε, ψηφοφοριών αυτό το σημείο, ως δεύτερο σημείο ή αν κάτι μπορούσαμε να κάνουμε που θα δώσει χρόνο ε, στι ομάδες, θα κάνουμε ως τελευταίο σημείο, θα έχουμε ψηφοφορίες και θα εντάξουμε αυτό το σημείο. Μόνο που δεν μπορώ να σας πω ακριβώς σε ποια ώρα θα γίνει αυτό, ποια ώρα θα το κάνουμε. Είναι μικρό πρόβλημα αυτό. Πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό είναι ένας κίνδυνος που υπάρχει. Είναι επισφαλής η κατάσταση. Αλλά θα ήταν δίκαιο και σωστό να έχουμε χρόνο οι συνάδελφοι και οι ομαδες μια μια-δυο ώρες να το δούνε το θέμα, να συζητήσουν μεταξύ του. Άλλε δυνατότητε δεν βλέπω να υπάρχουν. Εντάξει. Ή η τρίτη εναλλακτική λύση θα ήταν το μεσημέρι, το, την απογευματινή μα συνεδρίαση ως πρώτο σημείο να το είχαμε. Θα έχουμε και να φιλοξενούμε τον κύριο Έτιγκερ, δεν θα θέλαμε να ψηφίσουμε πιο πριν, αλλά και θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ο κύριος Βόμποντα όμω ζήτησε πάλι τον λόγο. Πρόεδρε, θα παρακαλούσα ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο να προβλέψουμε, όπως είπατε στο τέλος, χωρίς συζήτηση. Μία ώρα στην οποία θα γίνει ψηφοφορία, μόνο η ψηφοφορία. Πρόεδρος, επαναλαμβάνω την πρόταση. Ξέρω ότι δεν είναι απλό να το κάνει κανείς αυτό. Παρακαλώ όμως να είσαστε όλοι ακριβώς την ώρα σας. Στις 3 η ώρα λοιπόν θα λέγαμε. Πρώτο σημείο, στην απογευματινή συνεδρίαση θα εγγράψουμε την ψήφιση για αυτό το ψήφισμα. Και έτσι λοιπόν θα υπάρχει χρόνο να το συζητήσετε, να προβληματιστούμε και να δούμε. Θα ψηφίσουμε όμω στι τρει, Τελεία και παύλα. Γιατί δεν θέλω να αφήσω το φιλοξενούμενο να περιμένει. Έχουμε και ένα σημείο. εντάξει. Πώ είπατε εσεί. Uh, Μα μισό λεπτό χρειάζεται όλο και όλο. Είναι υπέρ ή κατά. Στι η ώρα θα το κάνουμε όμω, εντάξει. Λοιπόν, στι τρει, τελείωσε. Θα αλλάξει η ημερήσια διάταξη, το λέμε αυτό. Στις 3 η ώρα λοιπόν θα έχουμε ψηφοφορία για το θέμα αυτού του ψηφίσματος. Και μόνο θα ψηφίσουμε, τελείωσε, δεν θα υπάρχει συζήτηση. Κυρία Μαντουρέν, παρακαλώ. Κοιτάξτε πρόεδρε, οι μεγάλες ομάδες έχουμε περισσότερα προβλήματα για να έρθουμε σε επαφή με όλους από ότι οι μικρές ομάδες που με ίσως κάποιο τηλεφώνημα μπορούν να τα επιλύσουν για το, τις 3 το απόγευμα δεν θα γινόταν στα τέλη της απογευματινής συνεδρίασης ή τουλάχιστον στις 4 ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο διότι υπάρχουν πολλοί που πρέπει να έρθουμε σε επαφή δεν υπάρχει πρόβλημα να ψηφίσουμε μετά από την παρουσία του κυρίου Έτιγκερ εντάξει μετά την παρουσία του παρουσίαση του κυρίου Έτιγκερ να ψηφίσουμε Πρόεδρος, εντάξει, καλώ. Η γραμματεία είπε καλύτερα θα ήταν σήμερα το πρωί να το κάναμε, γιατί πρέπει να μεταφραστεί, να περάσει από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Να πούμε τρεις η ώρα, εντάξει, τρεις. Τρεις παρακαλώ, να είσαστε όλοι παρόντες. Συμφωνείτε, εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Είναι οι ψηφοφορίες αυτό για την έκθεση της κυρίας Μπαντιάη Κουτσέτ. Έχετε τα έγγραφα, τα χαρτιά μπροστά σας. Τις κάρτες σας τις έχετε, εντάξει. Μια στιγμή. Να βάλουμε την κάρτα στη συσκευή. Και αν συμφωνείτε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες τώρα. Wir machen es äh, immer Λοιπόν, με τον κατάλογο θα προχωρήσουμε όπως πάντα. Συμφωνείτε, πρέπει να προσέξουμε καλά-καλά να δούμε ποιες αλλαγές έχουμε. Η πρώτη ψηφοφορία, τροπολογία 41. 41 υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 1. Ποιοι είναι υπέρ. Μια, ένα, ένα λεπτό. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Διαδικαστικό, κύριος Γκασπάρη, παρακαλώ. Αξιότιμε πρόεδρε, θα έλεγα στη σημερινή ψηφοφορία έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Κάπως πρέπει οι γραμματεία της Επιτροπής ΙΤΟ ε, και Ίντερ δεν υπήρξε σωστό συντανισμό μεταξύ αυτών των γραμματιών, διότι στον κατάλογο ψηφοφορία λείπουν όλε οι τροπολογίε που αφορούν τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Ίντερ. Και γι' αυτό η ερώτησή μου προ την Επιτροπή Ήτρε, στη γραμματεία τη Επιτροπή Ήτρε, πώ θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Το ξαναλέω, λείπουν στον κατάλογο ψηφοφοριών οι τροπολογίε τη Επιτροπή ε, Ήτρε. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε μια γνωμοδότηση μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Πώ προτείνει να λυθεί αυτό το πρόβλημα η γραμματεία δεν μπορώ να απαντήσω. Δίνω τη σκητάρη στη γραμματεία. Μπορεί να απαντήσει. Ε, Έμβαση χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρος, εντάξει κύριε Κασπάρη, κυρίε και κύριοι, λέει η γραμματεία ότι σήμερα για πρώτη φορά πήραν στα χέρια τους τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε. Έχει, τυπωθεί, έχει ανατυπωθεί στα χέρια όλων σας, πράγμα που αληθεύει είναι εδώ παρούσα αλλά κανένας δεν θα είναι σε θέση τώρα να εντάξει αυτές τις προτάσεις στον πίνακα ψηφοφοριών. Οι κριτικοί επικρίσεις που ασκήθηκαν είναι ε, σωστές. Δεν μπορούμε να το αποσαφηνίσουμε. Δεν έχω και όρεξη να αποσαφηνιστεί σε βάθος. Τώρα ήρθαν τα έγγραφα αυτά. Δεν μπορούσαν ε, να ενταχθούν στον κατάλογο ψηφοφορία. Πάει αυτό. Ή λοιπόν θα αναβάλουμε την ψηφοφορία ή θα ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Υπάρχουν ενστάσει να μην ψηφίσουμε τώρα να το αναβάλουμε αν θέλετε. Διαφορετικά θα ψηφίσουμε. Και παρακαλώ, ναι εντάξει, είναι, θα έλεγα ανέσχυντο μεν, αλλά παρακαλώ να δείτε αυτή τη γνωμοδότηση μετά. Εσείς παρακαλώ. Αν παίρνουμε σαν σοβαρά το έργο κοινοβουλευτικών επιτροπών, δεν είμαι σε θέση, χωρίς να έχω δει αυτά τα θέματα πιο πριν, να ψηφίσω για αυτά. Είναι σημαντικό ποιε είναι οι απόψει αυτή τη κοινοβουλευτική επιτροπή μέσα από τη γνωμοδότησή τη. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε αυτά. Εσεί κύριε Τούρμε. Uh, Κοιτάξτε, αν ε, η γραμματεία της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ μπορεί να μας στείλει τα στοιχεία αυτά εγκαίρως, τότε δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσουμε τη δικασία. Αν δεν μπορούμε όμως να ψηφίσουμε, τότε μάλλον θα πρέπει να ψηφίσουμε αν το αποφασίσετε εσείς κύριε Πρόεδρε μόνο. Εντάξει, σύντομα. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, πρέπει να συζητήσουμε κύριε Πολύ γοργά θα το κάνουμε. Μπορούν να ξανακατατεθούν στην Ολομέλεια, αγαπητέ κυρίε ε, Κασπάρη, να μην χαθούν αυτέ οι τροπολογίε. Αλλά μην αναβάλουμε την ψηφοφορία για σήμερα. Λοιπόν, είχαμε μία τοποθέτηση υπέρ, υπέρ τη αναβολή, έτσι κατανόησα. Υπάρχουν άλλοι που λένε να μην αναβάλουμε, να ψηφίσουμε. Λυπούμε, πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε το θέμα. Αν θα αναβληθεί η ψηφοφορία ή όχι. Ποιοι είναι υπέρ τη αναβολή. Να σηκώσετε το χέρι σα. Υπέρ τη αναβολή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά τη αναβολή. Ευχαριστώ. Αποχές. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να ψηφίσουμε. Είναι θλιβερό αυτό βέβαια και παρακαλώ να μεριμνήσουμε σε συνολομέλεια να είναι διαθέσιμες οι τροπολογίες. Συμβιβασμό 1 τον διευθετήσαμε. Περνάμε στην Γιούρι 1, νομικών υποθέσεων 1. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογία 1. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε στη 47 τροπολογία. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 48 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την τροπολογία 48 ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Παρακαλώ να βάλετε σε λειτουργία τη μηχανή για να ψηφίσουμε το μηχανισμό. Τι, δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί. Κάποιος μπορεί να ε, κοιτάξει τι γίνεται με τις, τις συσκευές. Λοιπόν, λειτουργεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τις 48 ηλεκτρονικά. Εντάξει, όλα καλά. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ λέγεται. Λοιπόν, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε, μάλιστα. Παρακαλώ, κυρία Εκ. Ναι, ούτε και σε μένα λέει, είχε ανάψει, δεν λειτουργούσε. Ένας μόνο υπάρχει εκεί, ε, ναι. 52-50. 55-52 λέγεται στον πρόεδρο τώρα. Ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 25 22. My God, was denn jetzt? What jetzt? We do it again. Τι θα κάνουμε τώρα. Also ich habe gedacht, die sagen mir die richtigen Zahlen. Νόμιζα θα μου λέγανε <laughs> τα σωσ, τους σωστούς αριθμούς, αλλά με, 50, με τους 50 δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Θα το επαναλάβουμε. Επαναλαμβάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και πάλι. Παρακαλώ. Zwei EPP δύο από το ΕΛΚ παραπάνω. Τι γίνεται εδώ, παρακαλώ να αφαιρεθούν δύο ψήφοι από το ΕΛΚ. ενταξει περα πέρας ψηφοφορία. Πολύ ωραία. 24-20 το αποτέλεσμα. Όλα εντάξει λοιπόν. Okay. Παρ' όλα αυτά εγκρίθηκε λοιπόν. Περνάμε στη 49 τροπολογία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Η 50 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. 51 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Η 52 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. 56 τώρα. Τροπολογία 56. Εντάξει. «56 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Γιούρι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 67. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίθηκε. Καταπίπτει. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίθηκε. 70. Να ελέγξουμε λέτε. Εντάξει. 69. Ψηφίζουμε την 69. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 70 υπέρ. Κατά. Να επαναλάβουμε. 70 όσοι είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. 71 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Καταπίπτει, καταπίπτει. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 76 υπέρ Α, συγγνώμη, 73, μάλιστα, 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 3, ίνκο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Γιούρι 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 5 Γιούρι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 γιούρι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 89 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε. 88. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε και αυτή. 8 ήμκο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 93 υπέρ, κατά, απόχες εγκρίθηκε και αυτή 94 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2 Γιούρι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Γιούρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 117 υπέρ κατά ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε 117 ψηφίζουμε την 117 έρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας ένας από το ΕΛΚ παραπάνω Δύο από το ΕΛΚ παραπάνω. Τώρα εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 118 τώρα. Όχι, 118 ναι τώρα. Υπέρ, παρακαλώ. 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 12 υπέρ, Καταπίπτει, όχι, καταπίπτει. Λοιπόν, συμβασμός 12, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τώρα καταπίπτουν πολλές τροπολογίες. Φτάμε στην 125, φτάνουμε, υπέρ, 125. Κατά, όχι την 125, τι λέτε. Σωστό είναι. 125 λοιπόν και πάλι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η κυρία Κοχμερίν. Διαδικαστικό. Συγγνώμη, πρέπει να επανέλθω στην 119. Είχαμε εγκρίνει την 88. Θα έπρεπε να ψηφίσουμε την 119 μετά. Αφορά την επόμενη. Αν όχι την 119 τότε να ψηφίζαμε την 4 ΙΜΚΟ. Το δεύτερο τμήμα. Έχει δίκιο. Έχετε δίκιο. Σωστό. Ωστόσο για το δεύτερο τμήμα μόνο έτσι. Να, ευτυχώς που πρόσεξε κάποιος. Ωραία. Λοιπόν, να επανέλθουμε σύντομα στο αίτημα της κυρίας Κοχμερίν. 119 τροπολογία. Δεύτερο τμήμα. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ του δευτέρου τμήματος. Κατά. Αποχές. Δεν υπήρξε πρόβλημα. Βλέπετε εγκρίθηκε. Η 14 τώρα. Σωστό. 14 ήμκο. Υπέρ. Κατά. Ε, επαναλαμβάνουμε. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 1 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 2 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στο 4 τώρα. <laughs> Υπέρ. Στην τροπολογία 4. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 8 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 8. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 8. τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. Περνάμε στην 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η α A ε. Γιούρι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλα εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 22 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Απορρίφθηκε, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, απορρίφθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η ΣΥ της Γιούρη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές και αυτή απορρίφθηκε. Και τώρα συμβιβασμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η D, Γιούρι, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 33 υπέρ κατά αποχές και αυτή θα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 40. Το κείμενο τώρα στο σύνολο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Εντάξει όλα καλά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Όλα εντάξει λοιπόν. Και τώρα πρέπει κάποιες προσθήκες να κάνουμε, πρόσθετες ψηφοφορίες. Ψηφοφορία 1 υπέρ. Τροπολογία 1 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα τελική ψηφοφορία έτσι όπως τροποποιήθηκε πάλι ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά όλα εντάξει πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα ομόφωνη έγκριση συγχαρητήρια προς την συντάκτρια. Και τώρα, <clears throat> όπως τροποποιήθηκε σε σχέση με το ψήφισμα, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, έτσι, και σε αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα. Και αυτή η ψηφοφορία ομόφωνα, ομόθυμα ε, έδωσε έγκριση. Ευχαριστώ. Πάει αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ θερμά. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Στις 3 η ώρα να είστε εδώ θα ψηφίσουμε στις 3 ακριβώς να το θυμηθείτε και ακριβώς την ώρα σας. Εντάξει. Περνάμε στο σημείο 5 λοιπόν τώρα. Πρόκειται για την ολοκλήρωση. Έχετε την ημερήσια διάταξη στα χέρια σας. Ολοκλήρωση της ε, ε, εσωτερικής αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν επιτρέπετε παρακαλώ οι συζητήσεις εκτός αίθουσας, λίγη ησυχία στην αίθουσα. Ε, κάποιοι θέλουν να συζητήσουν, κάποιοι άλλοι θέλουν να ακούσουν όμως. Λοιπόν, έξω από την αίθουσα οι συζητήσεις καλύτερα. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση έχουμε μια γνωμοδότηση στα χέρια μας του συναδέφου κ. Τσουκαλά. Δίνω τον λόγο στον αγαπητό συνάδελφο αμέσως και πάλι παράκληση όλες οι άλλες συζητήσεις έξω από την αίθουσα. Ησυχία στην αίθουσα παρακαλώ. Είχε τον λόγο κύριε Τσουκαλά παρακαλώ. Wow. E-commerce is a key 21st century marketplace. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πάρα πολύ σημαντική. The European digital single market. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, καθότι δίνει τη δυνατότητα σε 500 εκατομμύρια καταναλωτές να συγκρίνουν προϊόντα μεταξύ τους το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του συνολικού πωλήσεων λιανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από το 5% και θεωρείται ότι 140 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, μολονότι αυξάνεται σε εθνικό επίπεδο το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο υστερεί. Από το 2006 έως το 2008 το μερίδιο του συνόλου των καταναλωτών που έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά τουλάχιστον ένα αντικείμενο προϊόν μέσω του ίντερνετ αυξήθηκε από το 27% στο 33% ενώ το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει σταθερό στο 6 7%. Το 51% των λιανοπολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πουλούν μέσω του ίντερνετ. Παράλληλα όμως μόνο το 21% χρησιμοποιεί το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, μολονότι ήταν 29% το ποσοστό αυτό το 2006. Την περίοδο αυτή που τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό έντονη οικονομική πίεση, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, καταναλώνουν περισσότερο χρόνο συγκρίνοντας τα προϊόντα μεταξύ τους, ηλεκτρονικώς προσπαθώντας να βρουν τις χαμηλότερες τιμές. Όλο και περισσότεροι πολιτές περνάνε στο ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να καταφέρουν να πουλήσουν περισσότερα προϊόντα και να σώσουν σαστικά τα καταστήματά τους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μεταμορφώσει λοιπόν την ε, εσωτερική αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πειράσει πάρα πολύ τι τιμέ καθώ επίση και τη δυνατότητα σύγκριση των προϊόντων. Ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται φραγμοί που δημιουργούν ένα κατακαιρματισμένο ακόμα περιβάλλον όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δυστυχώ, η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη είναι αυτή μια εικονική αγορά για του πολιτέ εκείνου οι οποίοι πουλούν προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί κυρίω στην Κίνα και χρησιμοποιούν web servers και υπολογιστές που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα, που τρέχουν λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί στις ΗΠΑ μέσω συναλλαγών που εξασφαλίζονται μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλων των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιούνται κάρτες που έχουν δημιουργηθεί από εταιρείες των Ηνωμένων και τις οποίες διαχειρίζονται εταιρείε που έχουν ε, την έδρα τους στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Το μόνο ουσιαστικά ευρωπαϊκό στην όλη αυτή αλυσίδα είναι οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, κανονισμοί και φόροι. Και δυστυχώς το στοιχείο αυτό είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τα περισσότερα εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να φανταστείτε ότι έχω μια προστατευτική στάση, ακριβώς το αντίθετο. Προσπαθώ να κάνω το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο πολύ πιο απλό, πολύ πιο αποτελεσματικό, προκειμένου να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες όλων αυτών των χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καταφέρουν να απτυχθούν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου και προκειμένου ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν τον Ευρωπαίο καταναλωτή. για 350.000 περίπου λιανικούς πολιτές Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή μια συμφωνία που υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ακόμα πιο ασφαλές για τους πολίτες, πολιτές με συγχωρείτε, αυτούς. Δυστυχώ όμω υπάρχουν ακόμα κάποιες αδυναμίες και κάποια κενά όσον αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα απλό, ασφαλές, αξιόπιστο πλαίσιο για το ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο προκειμένου όλοι οι πολιτές και καταναλωτές Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να συμμετέχουν. Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώην Επίτροπος Κούνεβα ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολύ καλές μελέτες και ανακοινώσεις που περιγράφουν πολύ καλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο και προτείνονται συγκεκριμένα και λύσεις τόσο ιδιωτικό τομέα όσο και ενό των καταναλωτών συμφωνούν για τα σημεία αυτά τα οποία έχει τονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουν να γίνουν οι απαραίτητε αλλαγέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά διαθέσιμα μέσα προκειμένου να καταφέρει να ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να καταφέρει να έχουμε τις οδηγίες για τον αθέμητο ανταγωνισμό, για τις υπηρεσίες, για την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών και άλλα νομοθετικά μέσα. Το πρόβλημα όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς ότι έχουμε πάρα πολλά διαθέσιμα μέσα. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή περισσότερο και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους και θα το καταφέρουμε αυτό αν καταφέρουμε να έχουμε τελικά μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την Ευρώπη. Και καταλαβαίνετε ότι η ηλεκτρονική αγορά αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από ότι η ε, γραφειοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ηλεκτρονική αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να έχει μια κοινή και νέα θέση για την προώθηση της αγοράς αυτής. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα υποβάλουν πολλές επικοδομητικές προτάσεις προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο ισορροπημένο και σύντομο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έντσο έχει τον λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι εισηγητής, σκεώδης εισηγητής για την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών και ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τσουκαλά για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους από την καθήλυν αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή ΙΜΚΟ, και να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση τη Επιτροπή, το πρόβλημα με αυτού του είδου το εμπόριο, το εμπόριο έχει να κάνει με την έλλειψη εναρμόνιση στο επίπεδο τη εθνική νομοθεσία, των εθνικών νομοθεσιών δηλαδή. Την προστασία των καταναλωτών, του κανόνε σχετικά με τον ΦΠΑ, καθώ και τι πληρωμέ. Τι αυτόματε πληρωμέ. Έτσι λοιπόν κάποιοι από τους εμπορευόμενους στο διαδίκτυο ακολουθούν περιοριστική προσέγγιση, δηλαδή αρνούνται κάποιες συναλλαγές σε κάποια κάτι μέλη, κάτι που δυσκολεύει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Τώρα, λύσεις για να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό θα βρούμε σίγουρα και στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Συμφωνώ με τον εισηγητή μας αλλά και με την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΜΚΟ ως προς την τήρηση και την υλοποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες. Εκεί απευθύνεται έκκληση στα κρατημέλη για να δώσουν τέρμα στην διακριτική μεταχείριση από πλευράς κάποιων εμπορευμένων που αρνούνται να προβούν σε συναλλαγές ή ασκούν διακριτική μεταχείριση κατά των καταναλωτών ανάλογα με την εθνική τους προέλευση ή τη χώρα προέλευσής τους τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, η τη χωρα προελευσης του τελο παντων κατα τα αλλα η προταση για την ενιαία θηρίδα στην, στο κείμενο αυτό, ενιαία θηρίδα όπου όλοι οι εμπορευόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στο κράτο μέλος κατοικία τους, αυτή η διαδικασία απλούστευση τη διαδικασία ε, εγγραφής και δήλωση του ΦΠΑ στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η πρόταση λοιπόν περί ενίας θηρίδας νομίζω θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο λίγο πιο ευρύ. Θα πρέπει να κατονομαστεί μια εθνική αρχή, η οποία να έχει σκοπό ακριβώς να καταγράφει τις επιχειρήσεις και τους ε, ενδιαφερόμενους για να ασκήσουν αυτές τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει και μια διαδικτύωση αυτών των ευρωπαϊκών εθνικών αρχών σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε λοιπόν με την εναρμόνιση των εμπορικών δραστηριοτήτων, αυτών των εμπορευομένων και των παρεχόντων υπηρεσιών που θέλουν να έχουν δραστηριότητα διασυνοριακή. Έτσι θα υπάρχει ένα νομοθετικό και εμπορικό πλαίσιο ενιαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω ω προ την καταχώρηση, την εγγραφή των εμπορευομένων. Έπειτα, Ίσως ε, να πρέπει να αναθέσουμε στην Επιτροπή την ευθύνη να παρακολουθεί τις ε, κοινέ προδιαγραφές για την εξουσιοδότηση προκειμένου να μπορεί κανείς να ασκήσει τέτοιου δραστηριότητε. Ταυτόχρονα οι πελάτες, οι καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν εύκολη, διαρκή και δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες. Λόγου χάρη στο όνομα του ε, εμπορευομένου, τον αριθμό μητρώου με τον οποίο έχει καταγραφεί ή άλλες λεπτομέρειες όπως τις δαπάνες, ε, τι κέρδη έχει και ούτω καθεξής. Επίσης, νομίζω ότι τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε μια γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, πέραν της κάθε εθνικής γλώσσας. Και θα πρέπει να απαιτήσουμε και εξουσιοδότηση για αυτό το είδος τις εμπορικές συναλλαγές, Ιδίω όταν πρόκειται για μάρκε, λογότυπα και προϊόντα ποιότητα γνωστά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά για να λειτουργήσει εύρυθμα εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι καταναλωτέ να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στι υπηρεσίε που παρέχονται από του εμπορευομένου. Ω προ την καταβολή του ΦΠΑ, η Επιτροπή θα πρέπει στο μέλλον να εναρμονίσει του ειδικού φόρου κατανάλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτόν τον τομέα, τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για τις ε, online πληρωμές με πιστοτικές κάρτες ή άλλους τρόπους, θα πρέπει εδώ να υπάρξουν κανόνες ασφάλειας, πολύ απαιτητικοί. Θα πρέπει η Επιτροπή να προωθήσει κανόνες ασφάλειας για τις συναλλαγές που γίνονται με πιστοτικές κάρτες ε, κάρτες που να γίνονται αποδεκτές με τρόπο ομοιόμορφο και να χρησιμοποιούνται με τρόπο ομοιόμορφο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ε, κρατών μελών. Αλλά όχι μόνο να υπάρξει τέτοια εναρμόνιση, να αρθούν και οι φραγμοί που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, στις μέρες μας, ως προς τις πληρωμές με τις πιστωτικές κάρτες. Κάποιες πληρωμές, διευθετήσεις δεν γίνονται αποδεκτές από τις επιχειρήσεις ή από τους ίδιους τους εμπορευομένους. Οι τυποποιημένοι λοιπόν κανόνες είναι αναγκαίοι για να έχουμε ένα νέο σύστημα και επίσης για να προστατεύονται και τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο ομοιόμορφο. Θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε διακριτική μεταχείριση από πλευράς των εμπορευμένων που ενδεχομένως να ζητούν ε, περισσότερα έγγραφα, φωτοτυπία της ποσοτικής κάρτας να αποσταλεί με φάξ ή φωτοτυπίες ε, αντίγραφα της, του δελτίου ταυτότητας και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να προσέξει και την ανεξαρτησία κάποιων εγγράφων που χρησιμοποιούνται για αυτέ τι συναλλαγέ ε, σε περίπτωση που προέρχονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ε, οι περιπτώσει Mastercard και Visa. Κάποιε φορέ οι καταναλωτέ πρέπει να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό σε αυτέ τι εταιρείε. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να ορίσει ένα όριο 0,2% για τις προμήθειες που παίρνει η, κάρτα, η εταιρεία Visa για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Και αυτό για τους σκοπούς της βιώσιμης οικονομίας που θέλουμε να προωθήσουμε. Ξέρουμε ότι ο τραπεζικό τομέα σε αυτή την περίοδο τη χρηματοπιστωτική κρίση παρόλα αυτά πραγματοποιεί σημαντικότατα κέρδη. Και οι καταναλωτέ αλλά και οι εμπορευόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν αγώνα για την επιβίωσή του. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να μπορούν να ωφεληθούν από ένα σύστημα συναλλαγών στο διαδίκτυο με τραπεζικέ κάρτε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τι τράπεζε θα πρέπει να δώσει μια ευρωπαϊκή εναλλακτική στι περιπτώσει Visa και Mastercard ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην, στο ε, δομέα ακριβώ των ε, πληρωμών στο διαδίκτυο. Θα μπορούσε να υπάρχει λοιπόν ένας τέτοιο φορέας, ειδικά για την Ευρώπη. Τώρα για τους ιστοτόπους του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα πρέπει να δοθεί μια σχετική ελευθερία έκφραση στου εμπορευομένους για τη δυνατότητα πρόθεση και διαφήμιση των προϊόντων του. Και αυτό για να αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εμπορευομένων, αλλά να υπάρξει και η βελτίωση τη προσφορά, δεδομένη τη κρίση την οποία διανύουμε, αλλά και των ποσοστών ανεργία που βλέπουμε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά στον τομέα των διασυνοριακών συναλλαγών είναι μια μοναδική ευκαιρία για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ευρώπης. Θα πρέπει αυτά να τα δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Προς αυτό το σκοπό θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να προβλέψει ένα πρόγραμμα στήριξης των διασυνοριακών συναλλαγών, ιδίως για τους ανέργους, τους άνεργους πολίτες. Να δοθούν κίνητρα οικονομικά ώστε να μπορέσουν τα άτομα αυτά να αντιμετωπίσουν την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονταν. βρίσκονται. Θα μπορούσαμε να επιδοτήσουμε λόγου χάρη την αγορά λογισμικών ή hardware εξοπλισμού για να διευκολυνθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι η πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις δικές μας προτάσεις για να προωθηθεί περαιτέρω το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι προτάσεις σας και οι ιδέες σας είναι ευπρόσδεκτες. Οποιαδήποτε παρατήρηση είναι για μας αναγκαία, ιδίως από τον πρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοχμερίν, επόμενη, παρακαλώ. Ευχαριστώ θέρμα, Πρόεδρε. Πολλά ήδη αναφέρθηκαν και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, να επικεντρωθώ σε λίγα ουσιώδη στοιχεία. Αφενός είναι τώρα επιτέλους η χρονική στιγμή να ασχοληθούμε με το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η παλαιά ε, οδηγία είναι πλέον ξεπερασμένη. Έπρεπε να έχει γίνει αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να έχει επικαιροποιηθεί το πλαίσιο αυτό με μια έκθεση κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έγινε αυτό. Όμω τώρα οι κανόνες πρέπει να αλλάξουν, διότι πολλά έχουν γίνει και στη χώρα που ξέρω καλύτερα, τη Γερμανία. Η Γερμανία μεταξύ 2001 και 2009 στη Γερμανία ο αριθμός των ατόμων που online αγοράζουν κάνουν συναλλαγές από 12,9 εκατομμύρια αυξήθηκε ο αριθμός σε πάνω από 32 εκατομμύρια και υπάρχει λοιπόν λόγος, έχει υπερτριπλασιαστεί περίπου κιόλα. έτσι πολλά έχουν γίνει, πολλά τεκταίνονται και πρέπει πολλούς κανόνες να τους επανεξετάσουμε που μέχρι σήμερα είχαμε. Και αυτό δίνει έναυσμα εκείνοι που κάνουν συναλλαγές στο διαδίκτυο ή αγοράζουν στο διαδίκτυο να μην έχουν αρνητική διακριτική μεταχείριση έναντι των άλλων που αγοράζουν σε μαγαζιά αυτά τα εμπορεύματα και κάνουν τις συναλλαγές τους σε καταστήματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα αυτό το πλαίσιο να αλλάξει. Θέλουμε μια νομική εξίσωση μεταξύ του online εμπορίου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του εμπορίου που είναι μέχρι σήμερα συμβατό εμπόριο στα μαγαζιά, στα καταστήματα. Εξίσωση των συναλλαγών και μόνο εκείνο να μπορεί να πωλείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο ίντερνετ και μόνο εκείνοι να μπορούν ως έμποροι να δραστηριοποιούνται που έχουν και ένα ανοιχτό μαγαζί. Δηλαδή προϋπόθεση για το εμπόριο online προέρχεται από μια εποχή όπου τελείως διαφορετικοί κανόνες ε, λειτουργούσαν στην αγορά και τώρα δεν λειτουργούν πλέον και τώρα θα πρέπει να βασιστούμε στο ότι οι πελάτες με καλύτερες προσφορές και με καλύτερες πιο διαφανείς τιμές θα μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους και να αγοράζουν, να έχουν βελτιωμένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και οι έμποροι να εξισώνονται, να εξισώνονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ε, που έχουν οι άλλοι οι έμποροι του στο συμβατικό εμπόριο με καταστήματα και μαγαζιά και όλα αυτά να μπορούν να, εξε, ελεγχθούν και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να υποβάλει μια νέα ρύθμιση για αυτό το πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και επόμενος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος David Μέρ έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή για την πολύ επικοδομητική συμβολή τους, για τα επικοδομητικά του σχόλια. Κατά την άποψή μας το πρόβλημα είναι τεράστιο και πολύπλοκο. Όπως υπόθηκε έχουμε προβλήματα στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, του συστήματος πληρωμών, του φόρου προσθεμένης αξίας. Τι γίνεται με τα προϊόντα φτάνουν στο τέλος του βίου τους ε, κτλ. Πολύπλοκο λοιπόν ζήτημα, το οποίο καταλήγει όμως σε ένα απλό ζήτημα όσον αφορά τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Μελετώντας το ζήτημα αυτό βλέπουμε ότι σε περίπου 50-55% των περιπτώσεων οι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν μέχρι και 10% αν όχι περισσότερο αν αγόραζαν προϊόντα διασυνοριακά ακόμα και αν βάλουμε όλα τα μεταφορικά καθώς επίσης και τα έξοδα συσκευασία. Στο 6% των περιπτώσεων όπου ο καταναλωτής έχει προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο, συνάντησε προβλήματα. Η εταιρεία, για παράδειγμα, δεν αποφάσισε να του πουλήσει το προϊόν αυτό, το αρνήθηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πολύ δύσκολο, στην πράξη δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί και έχει επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και στα πλαίσια των κρατών μελών και ιδίω για τα μικρά κράτη-μέλη. Αν αγοράσει κανεί διασυνοριακά κάτι ηλεκτρονικά, μάλλον ενώ αυτό μπορεί να ισχύει σε μεγάλα κράτη-μέλη, σε μικρά κράτη-μέλη είναι φύση αδύνατο τις περισσότερες φορές. Δεν μπορεί να αγοράσει κανείς κάτι διασυνοριακά, ηλεκτρονικά. Και καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο τους πολίτες μας, πρέπει να τους δώσουμε περισσότερα ωφέλη, πρέπει να τους βοηθήσουμε να προασπιστούν τα δικαιώματά τους στα διασυνοριακά όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεωρούμε επίση ότι έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία μπροστά μα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια μικρή επιχείρηση η οποία κατασκευάζει ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, τα ζήτηση από τους Ευρωπαίους καταναλωτές διασυνοριακά. Είναι πολύ σημαντικό και για τις μικρές λοιπόν επιχειρήσεις να μπορούμε να έχουμε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού διασυνοριακού εμπορίου το οποίο θα είναι πιο απλό, πιο ομαλό. Είμαστε σε επαφή με την Επιτροπή ΙΜΚΟ και είμαστε σαφώ υπέρ όλων των προτάσεων που γίνονται στην γνωμοδότηση τη δική τη Επιτροπή, σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάναν ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομο για να μην ε, δυσχεράνω τη συζήτηση. Α δούμε τα πράγματα από την άλλη όμω πλευρά. Για ποιο λόγο το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν προχωράει, δεν σημειώνει πρόοδο, ενώ το εθνικό ηλεκτρονικό εμπόριο σημειώνει πρόοδο. Και αυτό γιατί συναντάμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάποιους κακούς εμπόρους. Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο θα πεθάνει από αυτούς οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να το σκοτώσουν ακριβώς επειδή δεν σέβονται το καταναλωτή, επειδή διατηρούν μια τέτοια στάση. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν έχουν ζητήσει τον λόγο άλλοι συνάδελφοι. Αναγγέλλω λοιπόν προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 5η 6η Μαΐου 12 το μεσημέρι. Οι συνάδελφοι έχουν συνεννοηθεί και συμφωνήσει από ό,τι φαίνεται γι' αυτό. Δεν υπάρχουν ενστάσει. Αυτό θα κάνουμε. Αυτή θα είναι η προθεσμία. Και ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και τώρα περνάμε στο σημείο 6. Διακυβέρνηση του διαδικτύου. Επόμενα βήματα. Η κυρία Σούζα Βάγνερ είναι η συγγήτρια από πλευρά μα. Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα υπάρχει εδώ μόνο. Η βιντεοδιάσκεψη με τους επαείοντες. Πρώτον, είχαμε προβλήματα με τη μετάφραση, με τις μεταφράσεις. Μετά όταν αναβάλαμε υπήρχαν τεχνικά προβλήματα για τη βίντεο, βίντεο διάσκεψη. Δεν μπορεί σήμερα να διεξαχθεί αυτή. Παρ' όλα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι θα έπρεπε να πάρουμε την ευκαιρία εσείς ε, κύριε Φρανσίσκο Σόσα Βάγνερ να παρουσιάσετε την έκθεση και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τους επαΐοντες ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε υστερότερα, γενέστερα αυτή την πλευρά. Θα το συζητήσουμε. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεσή σας. Κύριε Σούσα Βάγνερ, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, κύριε Σούσα Βάγνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα σήμερα να μπορώ εδώ να έχουμε μπροστά μας τα άτομα που έχουμε προσκαλέσει ως παίοντες για αυτή, αυτό το θέμα της διακυβέρνησης του διαδικτύου που είναι το θέμα της παρέμβασης και της δικής μου έκθεσης. Αυτή τη στιγμή όλοι οι κύριοι ευρωβουλευτές, γυναίκες και άντρες έχουν ήδη το κείμενο στα χέρια τους, το κείμενο του ψηφίσματος και γι' αυτό μπόρεσαν να γνωρίσουν περί τίνος πρόκειται. Έχει διανεμηθεί εδώ και κάποιες μέρες σε όλες τις γλώσσες, επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τώρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει πιστεύω εγώ είναι εκτός αν ο πρόεδρος δώσει εντολή ή αποφασίσει κάτι άλλο να ακούσουμε ακριβώς πρώτα τους επαΐοντες, τους πραγματογνώμονες με τη σειρά που η ίδια η Προεδρία θα επισημάνει. Αληθεύει, έχουμε πρόβλημα <clears throat> με την παρέμβαση όσον αφορά την βιντεοδιάσκεψη. Όμως, τι να γίνει. Αν δεν είναι δυνατόν να συνδεθούμε μέσω βιντεοδιασκέψης, τότε θα μπορέσουμε από πλευρά των επαϊόντων που είναι παρόντε να συζητήσουμε τι παρεμβάσει του. Να του ακούσουμε λοιπόν σύμφωνα με τι ενδείξει και με τη σειρά που θα καθορίσετε εσεί, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, εντάξει, ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο να ακούσουμε τι κυρίε και κυρίου εμπειρογνώμονε. Να παρακαλέσουμε να δώσουν μια σύντομη παρέμβαση, εισήγηση από πλευρά του, εκείνοι που είναι παρόντε και παρούσες. Ο κύριος Φρέντερικ Ντόγκ, αν βλέπω σωστά, είναι ο, ο πρώτος και του δίνω τον λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτέ, κύριε και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να συνεισφέρω στο έργο τη Επιτροπή Ήτρε. Και ιδίως αυτή την σημαντικότατη έκθεση για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Ένα ζήτημα ζωτική σημασία για την κοινωνία του διαδικτύου. Ελπίζουμε εδώ να έχουμε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, όπως έχει γίνει και σε άλλα φόρα για την διακυβέρνηση στο διαδίκτυο και σε άλλες αρμόδιες ομάδες. Ήθελα κατά πρώτον να περιγράψω το πρότυπο διαδικτύου που υποστηρίζουμε. Και επίσης τι εννοούμε με το σύστημα αυτό, το τοπίο του ίντερνετ που πρέπει να διαμορφωθεί. Θεωρώ τις ενίες αυτές ε, σημαντικές για να αναπτύξουμε το διαδίκτυο. Η εφιέλων του διαδικτύου βασίζεται στην αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική του, που στηρίζεται στο γεγονός ότι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ή να δημιουργήσει κιόλας τον εξοπλισμό, το λογισμικό, τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να γίνει μια πλατφόρμα δημιουργίας και καινοτομίας είναι πολύ μεγάλη σημασία ε, να έχουμε μηχανισμού διακυβέρνηση του διαδικτύου τέτοια ε, ε, οικοδόμηση που να επιτρέπουν την διαφάνεια, τη συμμετοχή όλων, την κατανομή ευθυνών και αυτό για όλους τους σκοπούς ανάπτυξης του διαδικτύου. Αυτό το ονομάζουμε το πρότυπο ανάπτυξης του διαδικτύου. Και πιστεύουμε ότι αυτό το πρότυπο θα έχει συνέπειες σε, όλε, σε όλες τις που αφορούν τον άνθρωπο και χρήστη του ίντερνετ. Οι θεσμικές αλλαγές φαίνονται και στο επίπεδο του ΟΗΕ, στο Φόρουμ Διακυβέρνησης του ίντερνετ. Το IGF επιτρέπει την ανοιχτή, διαφανή και γεμάτη συμμετοχή, γεμάτο συμμετοχή μάλλον διάλογο για θέματα του διαδικτύου και επιτρέπει και την απομάκρυνση από παραδοσιακά και παροχημένα μοντέλα. Πράγματι, η IGF ή η αντίστοιχη ευρωπαϊκή πλατφόρμα είναι χρήσιμα φόρουμ στα οποία οι χώρες, τα κράτη-μέλη μπορούν ε, ισότιμα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να προβούν σε διαπραγματεύσεις και συνεννοήσεις. Η αξία του προτύπου αυτού έχει αναγνωριστεί πλήρως και από τον ΟΣΑ και ζητείται όλο και περισσότερο αποκεντρωμένη προσέγγιση στο διαδίκτυο, καθώς και προώθηση της ε, οικονομίας του διαδικτύου. Υπάρχουν μεγάλα παραδείγματα της σωστής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επιτρέπουν τη βελτίωση, αλλά ακόμη πιο συναρπαστικό είναι το πρότυπο του διαδικτύου, όπως έχει προταθεί από τα διάφορα φόρουμ και τις ομάδες που συζητούν για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πρότυπο, το μοντέλο του διαδικτύου. Πρώτον, ότι είναι ένα δίκτυο δεκάδων χιλιάδων επιμέρους δικτύων με κατανομή των ευθυνών. Δεύτερο, λειτουργεί λόγω της ε, συνεισφορά πολλών ευρωπαϊκών φορέων με διαφορετικό ιστορικό, όπως των ερευνητών, της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών και των ε, αξιωματούχων κυβερνήσεων. Αυτά είναι καθοριστική σημασία για την επιτυχία του διαδικτύου. Τρίτον, η ανάπτυξη του διαδικτύου βασίζεται στα ανοιχτά πρότυπα, τα οποία ε, αναπτύσσονται και κατανέμονται με τρόπο ανοιχτό. Έπειτα, το πρότυπο του διαδικτύου βασίζεται στην καθοριστική αρχή, όπως η αρχή του τελικού χρήστη που πολλές φορές μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε εντυπωσιακές και πολύ χρήσιμες εφαρμογές. Πολύ σύντομα το μοντέλο αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο και πολύ καινοτόμο πρότυπο με σκοπό την εύχρηστη αξιοποίηση του διαδικτύου. Στο οικοσύστημα του ίντερνετ όπως το έχουμε ονομάσει υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα διακυβέρνησης αυτού του μοντέλου. Έτσι περνάμε στο δεύτερο σημείο που ήθελα να αναπτύξω, το οικοσύστημα του διαδικτύου. Το οικοσύστημα του διαδικτύου είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε ένα περιβάλλον, ένα τοπίο περιβαλλόντων και κοινοτήτων, τα οποία είναι αλληλένδετα και μαζί αναπτύσσουν τεχνολογίες και εφαρμογέ που σκοπό έχουν να βελτιώσουν γενικότερα τη χρήση του διαδικτύου. Οι οργανώσεις αυτές μοιράζονται κοινέ αξίες για την ανοιχτή ανάπτυξη, την ελεύθερη ανάπτυξη του ίντερνετ. Οργανώσεις λοιπόν ε, τέτοιες είναι οι φορείς τεχνικής ανάπτυξης όπως η IGF, η Task Force για τη μηχανική του ίντερνετ και το Παγκόσμιο Consortium. Έπειτα για τις δυνατότητες του ίντερνετ έχουμε την ICAN ή τις ε, επιμέρους περιφερειακές ομάδες για το διαδίκτυο και άλλες ομάδες εγγραφής. Τρίτον, εταιρείες που παρέχουν υποδομές ε, για το διαδίκτυο όπως προμηθευτές, ε, παρέχοντες ε, υπηρεσίες και φόρουμ ανταλλαγής. Έπειτα οι χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να επικοινωνούν μεταξύ τους και παρέχουν και άλλες υπηρεσίες όπως το καινοτόμο λογισμικό ή και άλλες υπηρεσίες. Και πέμπτον, οργανώσεις που παρέχουν εφαρμογές και επιτρέπουν την οικοδόμηση δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και την πρόθεση των ε, εφαρμογών και των χρήσεων του ίντερνετ, όπως οι πολυμερείς, οι τοπικές, οι περιφερειακές, οι κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς. Θα ήθελα τώρα να θίξω ένα από τα θέματα που είναι ζωτική σημασία και στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στην έκθεση του κυρίου Βάγκνερ και να σταθώ στο θέμα της ICANN. Όπως θα βλέπετε από την περιγραφή του οικοσυστήματος του διαδικτύου, η ICAN είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στο οικοσύστημα αυτό. Αλλά να θυμόμαστε τι ήταν, ποια ήταν η εντολή της ICAN. Κυρίως να αναπτύξει τεχνικές ε, λειτουργίες. Αρκετά αυστηρός μάλιστα. Ως φορέας δεν είναι ο βασικός οργανισμός διακυβέρνησης του διαδικτύου, ούτως ή άλλως. Η κοινωνία του διαδικτύου πιστεύει ότι η ICAN είναι κάτι σαν εργαστήριο που επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία του συστήματος. Πρέπει η ICAN να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού και αυτό είναι ο βασικό τη στόχο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι ένα πρότυπο καλή διακυβέρνηση η ICAN. Σημαίνει ότι οι εξή βασικέ αρχέ πρέπει να είναι γνωστέ και να εφαρμόζονται. Πρώτα απ' όλα η διαφάνεια, δηλαδή η βελτίωση και συνεχής ανάπτυξη της έγκαιρης πληροφόρησης, οι πολυμερείς ε, διελτουργικότητες και η πλήρης διαφάνεια για τη λήψη αποφάσεων και της ε, λογιστικής βάσης της οποίας ελήφθησαν οι αποφάσεις. Έπειτα η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Τρίτον, αποδεκτικά στοιχεία για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τέταρτον, διάλογος με συμμετοχή είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το μοντέλο καλής διακυβέρνησης σημαίνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνομιλούν και εργάζονται μαζί ταυτόχρονα για τα ίδια ζητήματα που απασχολούν όλους προκειμένου να πετύχουν κοινή πρόοδο. Άλλα σημαντικά ζητήματα είναι το ζήτημα του υπόλογου και η ICAN έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι πολύ σημαντική για τέτοια ζητήματα υπολόγου. Και βεβαίω χρειάζονται, χρειάζεται ανταπόκριση και αντιδράσεις για το πώ λειτουργούν όλα αυτά, καθώ και ένα σύστημα διαδικασία, μια διαδικασία επίλυση των διαφορών. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει δει και η Αμερικανική κυβέρνηση και η ICAN στην ε, δήλωση των ε, δεσμεύσεών τους αλλά να είμαστε σαφεί. Το να επιτυχάνουμε τους στόχους και να παραμένουμε στη δήλωση των δεσμεύσεών μας θα είναι ήδη ένα βήμα πρόοδου, αλλά ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων θα είναι αυτός. Τα μέλη της κοινωνίας του διαδικτύου μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της ICAN μέσω των συμβουλευτικών φορέων και των υποστηρικτικών ομάδων και θα μπορούσαν το ίδιο να κάνουν και οι κυβερνήσει Εν είδη συμπεράσματο να θυμίσω τρία βασικά στοιχεία της παρέμβασής μου σήμερα. Πρώτον, στο οικοσύστημα του διαδικτύου η ICAN είναι σημαντικός φορέας αλλά δεν είναι και ο μόνος, ούτε ο πιο σημαντικός φορέας διακυβέρνησης. Δεύτερον, είμαστε πεπισμένοι ότι η οδήποτε θέμα έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, θα πρέπει να απειλείται κατά τρόπο συνεπή με το πρότυπο του διαδικτύου που έχουμε αναπτύξει. Δηλαδή, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της συμμετοχής, της συνεργατικής δέσμευσης και της ανοιχτής προσέγγισης. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωκοινοβούλιο έχουν μεγάλη ιστορία προώθησης του ανοιχτού προτύπου διακυβέρνησης. Το Ευρωκοινοβούλιο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εθνικές συζητήσεις για την ανάγκη το διαδίκτυο όπως θα δημιουργηθεί να είναι ανοιχτό και φιλικό προς το χρήστη. Νομίζω ότι η τωρινή συζήτηση αποδεικνύει ακριβώς την ίδια δέσμευση του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντική. Σήμερα η κοινωνία του διαδικτύου αντιμετωπίζει πολλές σημαντικές προκλήσεις και στην Ευρώπη. Οι προκλήσεις αυτές χρειάζονται μία ε, απάντηση τολμηρή από όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε το διαδίκτυο που θα δημιουργήσουμε να επιτρέπει ανοιχτή πρόσβαση, διαφάνεια και συμμετοχή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Επόμενος, ο κύριος Κιάν Κλίντς παρακαλώ. Πρέσβης. Χαίρομαι που είσαστε παρόν και προσβλέπουμε στις πληροφορίες και τη δική σας πείρα που θα μας παρουσιάσετε. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Thank thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σας για την σημερινή πρόσκληση, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω τις δικές μου απόψεις. Θα πάρω το λόγο βάσει της αρμοδιότητάς μου. Δεν εκφράζω αυτή τη στιγμή καμία κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι είμαι απόλυτα υπεύθυνος προσωπικά για οτιδήποτε πω και στηρίζω προφανώς τα λεγόμενά μου. Μου ζητήθηκε να αφαιρθώ σε τρία ζητήματα. Ένα από αυτά, το πρώτο, είναι η ICAN, η λογοδοσία της ICAN και η διαφάνεια για την ICAN. Προκειμένου να σας δείξω ότι πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό, πρέπει να σας πω ότι η ICAN δημιουργήθηκε το 1998 στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα με τη συμβολή πολλών ενδιαφερομένων και με τη συμμετοχή κυβερνήσεων που έχουν συμβουλευτικό καθεστώς. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα για το ρόλο που παίζουν οι κυβερνήσεις στην ICAN. Η ICAN, με άλλα λόγια, δημιουργήθηκε ως οργάνωση όταν ε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε εξωτερικούς συνεργάτες την διαχείριση και το συντονισμό των ε, συστημάτων ε, ίντερνετ ως νέα συσταθήσα οργάνωση, η ICAN, είχε μια πολύ αυστηρή υποπτία από την Αμερικανική κυβέρνηση μέσω ενός μνημονίου κατανόησης που είχε ισχύει από το 2006 και μετά και σύμφωνα με το οποίο επιβαλόταν στην ICAN από την Αμερικανική κυβέρνηση να υποβάλει κάθε χρόνο εκθέσεις, αναφορές με βάση τις επιδόσεις της. Στη συνέχεια, συμφωνία για το κοινό έργο JPA υπεγράφει για περίοδο τριών ετών και αυτό αποτέλεσε σημαντικό βήμα, σημαντική πρόοδο μετά το μνημόνιο κατανόηση στη συνεργασία που είχε η ICAN με την Αμερικανική κυβέρνηση. Η ICAN κατά αυτόν τον τρόπο κατάφερε να απομακρυνθεί από την αυστηρή εποπτεία της Αμερικανικής κυβέρνησης και σύμφωνα με τη Συμφωνία για το Κοινό Έργο υπήρχε μόνο μία πλέον αξιολόγηση το χρόνο της, ε, ε, των επιδόσεων της ICAN. Όταν ε, έφτασε το τέλος η συμφωνία αυτή, η Αμερικανική κυβέρνηση και η ICAN υπέγραψαν μια νέα συμφωνία αορίστου χρόνου που δεν προβλέπει καμία ρήτρα εποπτείας Αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά τις δραστηριότητες της ICAN. Προβλέπεται ότι η ICAN θα υποβάλει μία πολυετή έκθεση όσον αφορά τις επιδόσεις της, για ζητήματα όπως η λογοδοσία και η διαφάνεια και για την πολιτική που ακολουθεί, για την ασφάλεια του διαδικτύου και για τον ανταγωνισμό και την επιλογή του καταναλωτή. Η ICAN ίδια ως οργάνωση έχει ε, εγκρίνει ένα νομικό πλαίσιο και κάποιες νομικές αρχές όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Το Φεβρουάριο του 2008 εγκρίθηκαν οι αρχές αυτές και προβλέπονται τρεις μορφές λογοδοσίας. Πρώτον, λογοδοσία όσον αφορά το δημόσιο περιβάλλον, τη στιγμή που παρέχει μία υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος και μία δεύτερα, δεύτερη εταιρική λογοδοσία, λογοδοσία ουσιαστικά προς τις ε, συμμετέχουσες ε, επιχειρήσεις, προς τον επιχειρηματικό κλάδο δηλαδή που συμμετέχει στην ICAN. Σε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο ή σε αυτές τις αρχές πλαίσιο αν θέλετε, ε, προβλέπεται μια συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμογής. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ανάμεσα στους συμβαλωμένους στην ICAN για τις επιδόσεις της ICAN ως προς τους στόχους αυτούς. και έχει συσταθεί και μία επιτροπή αναθεώρησης, αξιολόγησης που θα συνεδράσει αύριο και μεθαύριο με στόχο να αξιολογηθεί και να αναθεωρηθεί το επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας της ICAN. Τώρα, πώς επηρεάζει η Κυβερνητική Συμβουλευτική Επιτροπή την ICAN. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από 100 περίπου μέλη και από 12 περίπου παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων χωρών όπως οι ΗΠΑ, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Καναδάς, αλλά και η Ρωσία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Αίγυπτος, Νότιος Αφρική, Κένια και πολλές άλλες χώρες συμμετέχουν σε αυτή την Επιτροπή. Στόχος της Κυβερνητικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ICAN είναι να δώσει κάποιες κατευθύνσεις όσον αφορά ζητήματα δημόσιας πολιτικής για οποιοδήποτε ζήτημα ουσιαστικά συζητείται στα πλαίσια της ICAN. Η Συμβουλευτική αυτή Επιτροπή έχει ένα ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το καταστατικό της ICAN, καθεστώς το οποίο διαφοροποιείται από άλλες συμβουλευτικές επιτροπές και που προβλέπει ότι σε περίπτωση απόρριψη μιας συμβουλή που δίνει η κοινοβουλευτική αυτή επιτροπή, το Προεδρείο της ΆΙΚΑΝ θα πρέπει να δώσει εξηγήσει για ποιο λόγο δηλαδή απορρίπτει τη σύσταση την κυβερνητική αυτή συμβουλή. Η κυβερνητική αυτή συμβουλευτική επιτροπή που υπάρχει από την αρχή ουσιαστικά της ΆΙΚΑΝ έχει εγκρίνει αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση των ε, domain names σε ορισμένες χώρες, αρχές ε, όσον αφορά ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο, υπηρεσίες όσον αφορά την ε, εκχώρηση των αριθμών και των ονομάτων στα πλαίσια του ίντερνετ. Από το 2007 και μετά η ICANN συμμετέχει στην, ε, στην ε, έγκριση δημοσίων πολιτικών όσον αφορά το διαδίκτυο. Η ICAN είναι μία οργάνωση bottom-up όσον αφορά την κατάρτιση ε, κατευθυντήριων γραμμών. Πρόσφατα όμως αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της και αντί να συμβάλλει ουσιαστικά στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας, η συμβουλευτική αυτή επιτροπή έχει αρχίσει να παρέχει συμβουλές από την αρχή της διαδικασίας κατάρτισης πολιτικής. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχει καταφέρει να συμβάλλει πάρα πολύ στην κατάρτιση του International Domain Name. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις τώρα για την κυβερνητική αυτή συμβουλευτική επιτροπή στα πλαίσια της ICAN. Καταρχάς, δεν έχει τους απαραίτητους πόρου. Πολλές φορές οι εθνικές κυβερνήσεις δεν δίνουν τα απαραίτητα χρήματα προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η επιτροπή αυτή της ICAN. Επίσης, δεν υπάρχει κατάλληλη γραμματιακή υποστήριξη. Και το μοντέλο το οποίο ακολουθεί η γραμματεία τη Βουλευτική αυτή επιτροπή δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Η Επιτροπή αυτή επίσης προσπαθεί να δει ποιε είναι οι διαδικασίες που ακολουθεί και εργαζόμαστε με το Προεδρείο της ΆΙΚΑΝ αυτή τη στιγμή προκειμένου να καταφέρουμε να ορίσουμε το ρόλο της ΓΑΓ, της Κυβερνητικής Αυτής Επιτροπής, στα πλαίσια της ICAN και να δυναμώσουμε το ρόλο της Κυβερνητικής Αυτής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η διεργασία αυτή θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και θα υποβληθεί μια έκθεση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ICANN που θα γίνει στις Βρυξέλλες στα τέλη Ιουνίου. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ και στο ζήτημα του μέλλοντος της Σύμβασης Αϊάννα. Όσοι δεν γνωρίζετε, η Αϊάννα είναι η αρχή του διαδικτύου για την εκχώρηση αριθμών. Με άλλα λόγια, Πρόκειται για μία λειτουργία διατήρησης και συντήρησης της βάσης δεδομένων αριθμών του διαδικτύου. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία συμφωνία ανάμεσα στην ICAN, τις Ηνωμένε Πολιτείε και τις εταιρείες εκείνες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία αυτή. Υπάρχουν δύο σαστικά συμβάσεις. Μία ανάμεσα στην IANA και την ICAN και μια άλλη σύμβαση ανάμεσα στην ΑΙΑΝΑ και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η πρώτη σύμβαση ακολουθεί τις ομοσπονδιακές ρυθμίσεις των ΗΠΑ. Στη σύμβαση αυτή έχουμε κάποιες συγκεκριμένους παραμέτρους επιδόσεων και στόχων της ICAN όσον αφορά την αρχή του διαδικτύου για την εκχώρηση αριθμών. Η ΆΙΑΝΑ είναι πάρα πολύ σημαντική για την ICAN. ουσιαστικά είναι ο λόγος ύπαρξης, αν θέλετε, της ε, ICAN. Η Αιάννα πρέπει να βελτιώσει τις επιδόσεις της και πιο συγκεκριμένα έχουμε κάποιες ε, στατιστικές ε, διαθέσιμες στο, στην ισοσελίδα της ICAN όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να βελτιωθούν οι δραστηριότητες της ΑΙΑΝΑ που αυτή τη στιγμή γίνονται εκτός Καλιφόρνιας, ενώ στο παρελθόν γινόντουσαν στην Καλιφόρνια, και θέλουμε λοιπόν να λειτουργεί κατά τέτοιον τρόπο η αρχή του διαδικτύου για την εκχώρηση αριθμών, η ΑΙΑΝΑ, προκειμένου να επέλθουν κάποιες ε, βελτιώσεις και προκειμένου να επεμβαίνει λιγότερο ανθρώπινος παράγοντας στη δικασία λήψης αποφάσεων. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ε, η ICAN είναι απλώς συμβαλόμενος στη συμφωνία αυτή. Επομένως, στο μέλλον οι συμβάσεις ΑΙΑΝΑ δεν θα πρέπει να συζητώνται στα πλαίσια της ICAN, αλλά κυρίως με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην έκθεσή σας, ε, κύριε Πρόεδρε, στο σημείο 25 λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ICAN θα πρέπει να περιέχει κάποιους μηχανισμούς διμερούς λογοδοσίας και ότι καμία χώρα θα πρέπει να έχει ανώτερη θέση, αν θέλετε, στα πλαίσια της ΑΙΑΝΑ. Το ζήτημα βέβαια είναι πολύ πλοκό. Αν έχουμε στόχο να επαναδιαρθρώσουμε το σύστημα συμβάσεων της ΑΙΑΝΑ θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει διεθνής διμερής ή ε, πολυμερής λογοδοσία. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο καθεστώς λογοδοσίας αν δεν καταλαβαίνουμε τι εννοούμε με τον όρο αυτόν. Σε πολλές περιπτώσεις Έχουμε προσπαθήσει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μελλοντική σύμβαση της ΑΙΑΝΕ και δεν το έχουμε καταφέρει. Πρέπει μεταξύ μόνο καταρχάς να συμφωνήσουμε και συνέχεια να προτείνουμε το όραμα μας αυτό στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, να δούμε αν συνάδει το δικό μας όρο με το δικό τους και να δούμε τελικά ποια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση, η ΑΙΑΝΑ θα πρέπει να λειτουργεί μέσω μιας εταιρείας, ενός φορέα που να έχει διεθνή παρουσία και που να μπορεί να επηρεάζει διεθνώς ουσιαστικά την εξέλιξη των πραγμάτων. Η ΑΙΑΝΑ θα πρέπει να είναι μια οντότητα με διεθνή παρουσία και επιρροή. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, επιτρέψτε μου. Επόμενος κύριος Πόλγκαρ, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Είμαι διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία της Πληροφορίας και ασχολούμαστε με θέματα οπτικο- οπτικοακουστικά μέσω μαζικής ενημέρωσης και διαδικτύου και είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας για δύο συγκεκριμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας διοργάνωση, πώς εμείς δουλέψαμε ως τώρα και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που δουλεύουμε. Κατά πρώτα να πω, Πρόεδρε, ότι δεν θα πάω πολύ μακριά στο παρελθόν διότι η ICAN ιδρύθηκε το 1998 και το διαδίκτυο νομίζω έκτοτε έχει αλλάξει πολύ. Σήμερα το διαδίκτυο έχει γίνει μια ζωτική σημασία ε, λειτουργία παγκοσμίω. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαν καθόλου να λειτουργήσουν οι κοινωνίες μας. Και κύριε Σόσα Βάγκνερ, ο συγκητής του Κοινοβουλίου, ε, χρησιμοποίησατε έναν πολύ σωστό όρο ονομάζοντας το διαδίκτυο ένα δημόσιο κοινό αγαθό. Τώρα, πώς λειτουργούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την εξέλιξη του διαδικτύου και πώς έχει εξελιχθεί και η ίδια η Μόνο μία αναδρομή στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, κατά τις συζητήσεις μας με τα κράτη-μέλη, τους ενδιαφερομένους, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, συνειδητοποίησαμε ότι η εκπνοή της κοινή της συμφωνίας κοινού προγράμματος μάλλον που συνδέει την Αμερικανική κυβέρνηση με την ICAN όπως θα ανέπτυξε και ο πρέσβης Κάρκινς η εκπνοή λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου πέρσι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτό συνειδητοποιήσαμε. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε την ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που σήμερα έχετε στα χέρια σας διακυβέρνηση του διαδικτύου τα επόμενα βήματα. Επιτρέψτε μου να παραθέσω μόνο δύο λόγια από αυτήν την ανακοίνωση που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις που ανταλλάχθησαν μεταξύ ενδιαφερομένων μελών του Ευρωκοινοβουλίου κρατών μελών. Δύο όροι ήταν ε, χαρακτηριστικοί. Ένα, η παγκοσμιοποίηση του ίντερνετ έχει γίνει διεθνές αγαθό, κοινό αγαθό το διαδίκτυο και δεύτερη, δεύτερος όρος, το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει να λειτουργούμε προς όφελος των πολιτών. Αυτά είναι τα δύο καθοριστικά μηνύματα στην καρδιά αυτής της ανακοίνωσης. Έχουν υποθεί πολλά για την ICAN και Χρησιμοποιούμε την ICAN γιατί ακριβώς εκείνη επεξεργάζεται το DNS. Το DNS είναι η υποδομή που βρίσκεται στην καρδιά ολόκληρου του συστήματος του διαδικτύου. Όμως έχει γίνει περισσότερο τεχνικός ε, φορέας, διαχειριστής για το DNS, ε, ο, η ICAN. Και έχει γίνει και ε, υπεύθυνη για τις οργανώσεις που λειτουργούν στο διαδίκτυο και υπάρχει και η ανάλογη συμβουλευτική επιτροπή. Είναι πραγματικά το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και είναι και τεχνικός διαχειριστής της υποδομής βάσει της οποίας λειτουργεί το διαδίκτυο. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι είναι σημαντικό το ζήτημα της διακυβέρνησης του διαδικτύου να το ξαναδούμε στο πολιτικό επίπεδο πέρυσι, λόγω της μελλοντικής εκπνοής της συμφωνίας του κοινού Γι' αυτό και σας υποβάλαμε την ε, ανακοίνωση αυτή. Η Σουηδική Προεδρία μελέτησε την ανακοίνωση αυτή και συνειδητοποίησε ότι ο χρόνος είναι πολύ λίγος εφόσον εκείνη η συμφωνία πρόκειται να εκπνεύσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Πολύ γρήγορα λοιπόν η Σουηδική Προεδρία προώθησε το θέμα στο Συμβούλιο για να ετοιμαστούν κατευθυντήριες γραμμές. Όχι με τον επίσημη διαπραγματευτική εντολή, διότι η ΑΕΚ είναι ανεξάρτητο φορέα. Δεν μπορούμε στο θεσμικό δημοσιοπλαίσιο που διαθέτουμε να ε, διαθετήσουμε αυτό το περίεργο. Υπάρχουν εντολέ για διεθνεί διαπραγματεύσει, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία γι' αυτό, αλλά με διεθνεί οργανισμού ή φορεί. Αλλά η φορει αλλα η ICAN δεν είναι ούτε κράτο ούτε διεθνή οργανισμό. Είναι ιδιωτικό φορέα, ε, μη κερδοσκοπικό, υπό τον νόμο, την νομοθεσία τη πολιτεία τη Καλιφόρνια. Έτσι λοιπόν ετοιμάστηκαν κατευθυντήριες γραμμές και αυτό για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη της Τρόικα στην Ουάσιγκτον στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για να είμαι ακριβής, τέλη Αυγούστου πέρσι. Η Τρόικα, ως ήθιστε, το, από την Προεδρία, την ασκούσα Προεδρία, που ήταν η Σουηδική όπως προείπα, την ε, επερχόμενη Προεδρία, την τωρινή δηλαδή την Ισπανική, και την Επιτροπή που εκπροσωπείται από τον κύριο Φάμπιο Κολασάρτη, τον πρώην Γενικό μας Διευθυντή. Το μήνυμα που απεστάλλει μετά με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές του Συμβουλίου είναι ότι και εκείνοι εμπνεύστηκαν από την ανακοίνωση της Επιτροπής και το δικό μας μήνυμα ήταν διεθνοποίηση και κοινό συμφέρον, κοινό όφελος. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκε η ανακοίνωση και βάσει αυτών ε, η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Αμερικανικής Κυβέρνησης και ICAN επικροτήθηκε από την Επιτροπή ως ενδεχομένως θετικό βήμα πρόοδου. Η δήλωση δεσμεύσεων αναφέρει ρητός την ανάγκη να διασφαλίσει η ΑΕΚΑΝ ότι οι αποφάσεις τη είναι σύμφωνες με το δημόσιο συμφέρον και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ενδιαφερομένων. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη και ανάλυση των ε, επιπτώσεων των αποφάσεων θετικών ή αρνητικών στο κοινό. Αλλά αυτό δεν είναι απλώς μια δήλωση πίστης. Υπάρχει συγκεκριμένη εντολή για ομάδε αναθεώρηση. Οι ομάδε αυτές αναθεώρηση αποτελούνται από εθελοντές από όλο τον κόσμο. Δεν αναγνωρίζουμε λοιπόν απλώ την δημόσια, τον ρόλο που ασκεί μάλλον η ICAN στην χάραξη δημόσια πολιτική, αλλά και την παγκοσμιοποίηση του διαδικτύου. Οι ομάδε αυτέ αναθεώρηση έχουν ξεκινήσει το έργο του. Η πιο σημαντική είναι αυτή που ασχολείται με τη λογοδοσία και την διαφάνεια τη ICAN. Ο κύριος ε, Κάκλιν ανέφερε τις υπόλοιπες, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές, αλλά δεν θα επαναλάβω την απαρίθμηση αυτή. Το AOC λοιπόν το επεξεργαστήκαμε και μας ικανοποίησε ιδιαίτερα η ετοιμασία του. Είναι ίσως ένα θετικό βήμα προόδου, σκεφτήκαμε, αλλά ενώ μεταξύ τίποτε δεν συνέβη. Υπεγράφει στις 30 Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο τίποτε δεν έγινε. Ή τουλάχιστον δεν είχαμε εμεί καμία ένδειξη. Το ίδιο το Νοέμβριο. Οι προθεσμίε ήταν πολύ αυστηρέ και η πρώτη ομάδα αναθεώρησης έπρεπε να υποβάλει την πρώτη της έκθεση στο τέλος της φετινής χρονιάς. Αρχίσαμε κάπως λοιπόν να αγχωνόμαστε για αυτήν την πρώτη καθυστέρηση. Και συλλογικά αποστήλαμε το πρώτο σαφές μήνυμα. Πρώτον, μέχρι τον ΚΑΚ της Σεούλ στα τέλη της περασμένης χρονιάς και έπειτα μηνύματα στο IGF στο Σάρμελ Σέκ. Οι ευρωβουλευτές που παρέστησαν στη συνάντηση αυτή μας εξυπηρέτησαν ιδιαίτερα στο να είναι σαφή τα μηνύματά μας αυτά. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν έχουμε την πρώτη πρόταση για τη δημιουργία ομάδας αναθεώρησης. Η πρώτη τέτοια ομάδα συστάθηκε επιτέλους. Αποτελείται από 13 μέλη, 4 κυβερνητικά μέλη από την πλευρά τη συμβουλευτική των ε, κυβερνήσεων. Εκπροσωπούνται λοιπόν και οι κυβερνήσεις. Η γεωγραφική ισορροπία είναι λίγο πολύ σωστή. Διότι εκπροσωπούνται βεβαίω οι στο πρόσωπο του κ. Στρίτκλιν έναν αντιπρόεδρο της ΓΚΑΚ από την Αίγυπτο, την κυρία Ισμαέλ, ένα γενικό διευθυντή από Κινέζικο Υπουργείο και τον κύριο Κολασάντη, ο οποίος όπως είπα προηγουμένως συνταξιοδοτήθηκε από την αρχική του θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Γενικό Διευθυντή. Η σύνθεση της ομάδας λοιπόν είναι καλή αλλά πρέπει να αρχίσει και να δουλεύει ξεκίνησε και οι πρώτες συναντήσεις έγιναν όπως είπε και ο πρέσβης Κάρκιν στην αυτή την εβδομάδα μόλις. Σήμερα μάλιστα προβλεπόταν συνάντηση, γι' αυτό θα είχαμε και άλλους παρόντες, αν δεν υπήρχε συνάντηση αυτή, και ελπίζουμε η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί ομαλά ήδη έχει ξεκινήσει καλά. Υπήρχαν κάποιες διασκέψεις και θα υπάρξουν και κάποιες διαζώσεις συναντήσεις τον Ιουνίο πριν από τη συνάντηση της ΆΕΚΑΝ στις Βρυξέλλες. Τότε πραγματικά θα μπορούμε να αποτιμήσουμε τι πρόοδος έχει επιτελεστεί. Και αν πρόκειται να επιτευχθεί ο σκοπός των δηλώσεων για την λογοδοσία και τη διαφάνεια στο τέλος της χρονιάς. Λίγο πολύ έτσι έχουν πάει τα πράγματα ως τώρα, Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα λόγω και της δικής σας, ε, του δικού σας ενδιαφέροντος για το θέμα αυτό και φυσικά είναι σημαντική συμμετοχή των Αμερικανών. Να θυμίσω το πρόσφατα λόγια του κυρίου Στρίκλιν, που είναι υπεκεφαλής ε, της Αμερικανικής κυβέρνηση για τα θέματα οπτικοακουστικών και μέσων μαζική ενημέρωση. Ε, Λόγο που εκφωνήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 29 Απριλίου του 2009 μιλούσε για τα συστήματα του διαδικτύου στο 3,0. Λέει ότι η ICAN παραμένει ένας από τους σημαντικότερους φορείς στον κόσμο για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και από τη δική μας σκοπιά λέει, των Αμερικανών δηλαδή, είναι σκόπιμο οι κυβερνήσεις να συμμετέχουν στην ICAN επειδή είναι ζωτική σημασία η συμμετοχή τους ώστε οι αποφάσεις της ICAN αντικατοπτρίζουν το κοινό καλό. Αυτό είναι πραγματικά μια πραγματική αλλαγή στη στάση, την παραδοσιακή στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης προς την ICAN. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα, Πρόεδρε. Και για τα ενδεχόμενα βελτίωση. Να πω ότι μέχρι τώρα θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί. Όσο προχωρούμε προς τη συνάντηση της ICAN στις Βρυξέλλες του Ιουνίου, και τη συνάντηση του IGF στο Βίλνιους το Σεπτέμβριο, βλέπουμε παρόλα αυτά ότι η συνεργασία μας με το Ευρωκοινοβούλιο παραμένει εξαιρετική, πολύ καλή. Νομίζω οι βουλευτές εδώ θα συμφωνούν. Νομίζω η έκθεση του κυρίου Σόζα Βάγνερ φτάνει στην κατάλληλη στιγμή, διότι συμπίπτει με τη συνάντηση αυτή τη ΣΑΕΚΑΝ και τι σημαντικέ αποφάσει που θα πρέπει να ληφθούν εκεί για την λογοδοσία και το, τη διαφάνεια και του σκοπούς που επιδιώκουμε μέχρι το τέλο του χρόνου και βεβαίω μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη και πιο συστηματική συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου σε πρώτη φάση. Εμεί, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε απόλυτα ανοιχτοί στο να διαβρούμε, να εξεύρουμε μάλλον το σωστό τρόπο συνεργασία μαζί σα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ θερμά εγώ και βλέποντας τον χρόνο, το ρολόι, να επισημάνω ότι είχαμε συμφωνήσει κάθε επαΐων να έχει 5 έως 10 λεπτά στη διάθεσή του για να μας καλύψει ο χρόνος. Θα ήθελα όμως να μπορούν και οι συνάδελφοι να διατυπώσουν ερωτήσεις στη συνέχεια. Επόμενος, ο κύριος Μπράουν, παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας για να μιλήσω σήμερα για την διακυβέρνηση του ε, διαδικτύου. Όλο και περισσότερο η κοινότητά μας ε, βασίζεται σε αλλοσυνδεμένα συστήματα και στην ασφάλεια των συστημάτων αυτών. Πολύ σωστά ο κύριος Βάγνερ στην έκθεσή του λέει ότι θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμα συστήματα τα οποία είναι πιο ανθεκτικά, να έχουν τις κατάλληλες ασφαλείς υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, ιδίω μέσω του μεταρρυθμισμένου πακέτου μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, προκειμένου να παρέχεται ασφαλή συνεχής υπηρεσία σε όλους τους καταναλωτέ. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν αρχίσει να συζητούν ήδη τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φτάσουν σε ένα κοινό επίπεδο ασφάλεια στο διαδίκτυο με, με τι απαραίτητε ομάδε σε εθνικό επίπεδο που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια αυτή. Η ΕΝΗΣΑ θα πρέπει να παρέχει ένα φόρουμ για ανταλλαγή πληροφοριών και να υποστηρίζει τα λιγότερα ικανά κράτη-μέλη. Δεύτερον, θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο αποτελεσματικότητα τη ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία δηλαδή Δικτύων και τη Κοινωνία τη Πληροφορία, να τη δοθούν τα απαραίτητα μέσα και χρηματοδοτικά και θα πρέπει στα πλαίσια τη συνθήκη τη Λισαβόνα να μπορεί να λαμβάνει δράση και στα... στον τρίτο πυλώνα πλέον. Επίση, θα πρέπει ε, σημαντικοί τομείς του κλάδου να ρυθμιστούν περισσότερο. Θα πρέπει να έχουμε τις ε, απαραίτητες δομές όπως προσβλέπονται από το 144-2008 από την οδηγία αυτή του Συμβουλίου και θα πρέπει επίσης να έχουμε τα απαραίτητα utility systems για να ανταποκριθούμε αποκριθούμε στις ε, απαιτήσει ασφάλειας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών από τις υπηρεσίες ασφαλείας προς άλλους ενδιαφερομένους τομείς και θα πρέπει να ακολουθείται ο νόμος για την ανταγωνιστικότητα καθώς επίσης και νομοθεσίες που υπάρχουν για την πολιτική προμηθειών. Μια παράκληση κύριε Μπράουν. Οι διερμηνείς δυσκολεύονται με αυτό το ρυθμό. Λίγο πιο αργά παρακαλώ. Έχουν πρόβλημα να διερμηνεύσουν με τέτοιο ρυθμό, με τέτοια ταχύτητα. Λίγο πιο αργά παρακαλώ. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο και να καθοδηγηθεί, να οδηγηθεί με συγχωρείτε προς το επίπεδο της απόλυτης ασφάλειας με την συνεργασία διεθνών εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνεργασία των κρατών μελών και των Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποφασίσει ποιος θα, πώς θα διαρθρωθεί ο ηγετικός αυτός ρόλος. Αναφέρθηκα σε κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν την υποστήριξη της ICAN προκειμένου να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και ασφάλεια του συστήματος διεθνούς τομέα θα πρέπει σε διεθνή φόρουμ όπως την Ηνωμένα Έθνη, ο ΩΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να υπάρχει απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να έχουμε συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του διαδικτύου και επίσης να δούμε ποια θα είναι η ευθύνη σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας των web browsers applications. Επίσης, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει το ρόλο του προωθώντα θεμελιώδεις αξίες όπως ελευθερία της έκφρασης και ιδιωτική ζωή. Το σχέδιο έκθεσης προτείνει να αυξηθεί ο κανονισμός Ρώμη 2 προκειμένου να καλυφθούν και άλλοι τομείς. Αυτό είναι πολύ θετικό και είναι πολύ θετικό επίσης να καλυφθούν και οι διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν για προσφυγές σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πολύ προσεκτική όταν προτείνει, το Συμβούλιο με συγχωρείτε, όταν προτείνει συγκεκριμένη νομοθεσία για τους φορείς IP θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά θα ζημιώσουν ουσιαστικά την ε, διακυβέρνηση του διαδικτύου και ουσιαστικά θα προωθήσουν τα κράτη εκείνα τα οποία δεν συμμερίζονται τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το διαδίκτυο. Θα ευχαριστώ θερμά. Και συνεχίσουμε με τη σειρά, όπως προβλέπετε, στη συνέχεια. Ο κύριος Τσούκ, παρακαλώ. Έτσι προφέρετε, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη και το χρόνο που πιέζει, να είσαστε συντομότερος. Uh, uh, uh, Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για την ε, προσοχή σα. Θα ήθελα να αναπτύξω κάτι διαφορετικό. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε για την διακυβέρνηση του διαδικτύου. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η διακυβέρνηση αυτή θα τη χρειαστούμε και 10 χρόνια από σήμερα. Και ο στόχο δεν είναι να καλύψουμε μόνο την ανταλλαγή πληροφοριών και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά να δημιουργήσουμε και την κατάλληλη κουλτούρα στην κοινωνία για τι νέε μορφέ επικοινωνία μα. Η κοινωνία πλέον δεν ζει μόνο στο διάστημα μετά την βιομηχανική εποχή, αλλά και στη διασύνδεση όλων των ανθρώπων μεταξύ τους. Ζούμε σε μια μορφή κοινωνίας που θυμίζει διαφορετικά πρότυπα, όπως την αρχαία αθηνανική δημοκρατία. Και βρισκόμαστε και σε συνεχή εξέλιξη. Είναι λοιπόν σημαντικό να τα έχουμε αυτά κατά νου καθώς συζητούμε. Κάτι που ενδεχομένως να είναι αρνητικό είναι ότι χάνουμε την ε, δυνατότητα να έχουμε ως σημείο αναφοράς μία μόνο ευφυή προσέγγιση και ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα συλλογικά. Είναι σαν να αναπτύσσεται μια νέα μορφή ανθρώπου, ανθρώπου του, αστοανθρώπινου είδους και αυτό θα πρέπει να σκεφτούν οι κυβερνήσεις για τα παιδιά του σήμερα. Η γενιά του ίντερνετ σημαίνει ότι μπορεί να επηρεαστεί και ο εγκέφαλος ακόμα και ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκέφαλος των ανθρώπων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεαστούν οι επικοινωνίες από τις τεχνολογίες. Θα είναι ο άνθρωπος του αύριο ικανός για πολλά διαφορετικά πολλές διαφορετικές λειτουργίες ταυτόχρονα. Για τους ανθρώπους που είναι κατά των 10 βέβαια, ε, δεν είναι δυνατόν το ποσοστό του 30% που αναλογεί σε κάθε λειτουργία να τηρηθεί. Όμως, για αυτήν τη νέα γενιά πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι η διακυβέρνηση του διαδικτύου και πώς θα τους επηρεάσει. Πρέπει να σκεφτούμε πώς μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα σε μια πρώτη φάση η μάθηση δεν είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται όπως εμείς. Για αυτούς η μάθηση είναι παιχνίδι. Πώς νόμοι λοιπόν θα επηρεάσουν ε, την εκπαίδευση και τη μάθηση. Έπειτα οι νέοι δεν βλέπουν το σχολείο στο σημείο αναφοράς, το πιο σημαντικό τόπο στη ζωή τους. Είναι ένα σημείο που συναντούν τους φίλους τους. Διαζώσεις. Έτσι λοιπόν η αντίληψη τους δεν είναι τόσο γραμμική ή κειμενική όπως των ε, προηγουμένων γενεών ή στην εποχή της φωτογραφίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε τα διάφορα επίπεδα μάθησης, πώς περνάμε από το ένα στο άλλο και να αναγνωρίσουμε ότι οι πληροφορίες ανταλλάσσονται πολύ γρήγορα μέσω των τηλεοπτικών δικτύων, των διάβλων επικοινωνίας. Πρέπει να καθορίσουμε διάβλους ανταλλαγής πληροφορίας και χρήσιμων ε, γνώσεων που χρησιμοποιούν οι νέοι και επίσης τις διαδικασίες επεξεργασίας που θέτουν σε εφαρμογή. Μη ε, γραμμική σκέψη λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι διάφορα μέρη της πληροφορίας μπορούμε να τα δούμε ξεχωριστά και να τα ενώσουμε σε ένα σύνολο χρήσιμο. Αυτό επηρεάζει όμως όλη τη ζωή των νέων, όχι μόνο τη μάθηση. Μπορούν ε, σε μια να ερμηνεύσουν πολύ πιο εύκολα εικόνες, να περάσουν σε μια ταυτόχρονη ερμηνεία πολυμέσων και να αναπτύξουν διαφορετικές λειτουργίες. Αυτό πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει την ε, διακυβέρνηση και να δούμε πώς θα επηρεαστεί βεβαίως και ο ιδιωτικός βίος των πολιτών και των νέων. Νέες μορφές κατανόησης, ε, η εξερεύνηση των πληροφοριών, το σκάνινγκ, η χρήση πόρων από πολλές διαφορετικές πηγές. Οι ε, νέες λειτουργίες θα είναι κάτι που θα το χειρίζονται οι ίδιοι πλέον οι μαθητές και οι φοιτητές και όχι αυτοί που μαθαίνουν δηλαδή και όχι τόσο οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Στην δεκαετία του 80 ένα βιβλίο προέβλεπε ότι περνάμε από την εποχή της έκθεσης ή του κειμένου όπου σκεφτόμαστε πάρα πολύ τα πράγματα στην εποχή της show business. Κάτι που θυμίζει την Αμερική και το Las Vegas. Ποια είναι τώρα τα αποτελέσματα για την κριτική σκέψη και την ε, γνώση μας. Να σκεφτούμε, θα μπορούσαμε να θυμηθούμε τα σενάρια του George Orwell. Εδώ θα επιδείξω κάποιε από τις διαφάνειες. Αλλά ο πιο χαρακτηριστικός ε, χαρακτήρα είναι ο Huxley. Που μας θυμίζει ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε γίνει πλέον συνεχώς αγχωμένοι και σε αντιστάθμισμα αναζητούμε συνεχώς τη διασκέδαση. Τη δεκαετία του 80 είδαμε να φτάνουμε λίγο πολύ σε αυτή τη μορφή ανθρώπινου ανθρώπινης συμπεριφοράς που συνδέεται στενά με το διαδίκτυο. Τα οπτικά δεδομένα δεν επιτρέπουν την πολύ βαθιά επεξεργασία και κατανόηση και περισσότερο επιζητούν την ψυχαγωγία. Εάν λοιπόν συνδυάσουμε αυτήν τη νέα κουλτούρα με την διαδικτύωση στο ίντερνετ, πολλοί θεωρούν ότι εδώ έρχεται και το τέλος της μοναξιάς αυτού του συναισθήματος, αλλά νομίζουμε ότι η διασύνδεση της εποχής της διασημότητας με την εποχή της διαδικτύωσης μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα. Οι νέοι αντιμετωπίζουν πλέον διαφορετικά τον ε, αυτό τους όπως προβάλλεται προς τα έξω. Μπορούν εκατοντάδες άνθρωποι να σε δουν στο ίντερνετ, στο Twitter λόγου χάρη. Πώς λοιπόν θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αυτό είναι ένας άμεσος αντίκτυπος του διαδικτύου στους νέους. So, one uh, Ένα στοιχείο για τη διακυβέρνηση που με μου έκανε εντύπωση στην ε, ανακοίνωση είναι αυτά για τον ιδιωτικό βίο. Μου φαίνεται λίγο παροχημένη εδώ η προσέγγιση. Φαίνεται ότι οι έφηβοι στέλνουν 4.000 μηνύματα το μήνα. Αν κάνετε έναν υπολογισμό, σημαίνει ότι δεν περνούν περισσότερο από 5 λεπτά στο καθένα. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει ελαφρώς. Και πετώντας προς τα εδώ χθε το βράδυ, διάβασα ότι οι καταναλωτές 10 έως 18 ετών περνούν 10,7 ώρες την ημέρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά στην ουσία μιλάμε για ένα οκτάωρο επειδή κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα τα παιδιά αυτά. Δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε αυτά αν προσπαθήσουμε να τα ορίσουμε, ούτε θα μπορέσουμε να ορίσουμε τον ιδιωτικό βίο ε, για την γενιά των ανθρώπων που σήμερα είναι 10 ετών. Τι θα γίνεται δηλαδή σε 10 χρόνια από σήμερα που θα είναι 20. Εδώ επίσης επηρεάζεται και η ανθρώπινη σκέψη στον εγκέφαλο τον ίδιο. Στον επιστημονικό τομέα βλέπουμε ότι οι, ανα, επιστήμονες θα αλλάξουν και το, πρώτο, το σχέδιο του εγκεφάλου. Ε, διότι οι ανάγκες μας καθορίζονται από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε ενώ υπήρχε η λειτουργία της μίμησης προηγουμένως και ενώ οι ψυχολόγοι λένε ότι λειτουργούμε με βάση τις προσκολήσεις μας, βλέπουμε να επηρεάζεται και το σχέδιο του εγκεφάλου που έχει βαθιά κοινωνική δομή. Όλα αυτά τα αντικατοπτρίζονται στον εγκέφαλο οι επιρροέ της κοινωνίας του διαδικτύου. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει πολύ σκεπτόμενη την ε, διακυβέρνηση του διαδικτύου. Όμως σκεφτείτε ότι έτσι κι αλλιώ αυτά που βλέπουμε σήμερα σε 10 χρόνια από τώρα ριζοσπαστικά θα έχουν αλλάξει. Το διαδίκτυο δεν θα είναι μόνο ανταλλαγή πληροφοριών ή ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά θα είναι ανταλλαγή εμπειριών. Όλη μας η εμπειρία θα περνάει από το διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάρα πολλές πληροφορίες μας δώσατε, πληθώρα πληροφοριών επιπρόσθετα. Πράγμα το οποίο είναι επικοδομητικό για μας. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία κάποιες παρατηρήσεις ή κάποιες ερωτήσεις να διατυπώσουμε και να επικεντρωθούμε στους συναδέρφους. Να δούμε. Η ε, κυρία Τράουτμαν πρώτη, παρακαλώ. Euh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον ε, συναδελφό μας Βάγνερ για την υψίστη ποιότητα της ε, γνωμοδότησής του και να ευχαριστήσω και όλους τους κοιόδης ηγητές που συνέβαλαν στην εργασία αυτή. Να ευχαριστήσω επίσης και τους εμπειρογνώμονες που είναι εδώ πέρα σήμερα μαζί μας, οι οποίοι μας εξήγησαν με τρόπο ιδιαίτερα διεξοδικό πώς λειτουργούν αυτά τα περίφημα review panels, αυτά τα panel αναθεώρησης και αξιολόγησης μάθαμε στην πράξη πώς λειτουργούν και θεωρώ ότι η γνώση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί από την ποιότητα των εκθέσεων αυτών θα καταφέρουμε να επιβεβαιώσουμε στη συνέχεια την ποιότητα των δεσμεύσεων της ICAN και τις ε, περαιτέρω αρμοδιότητες της ICAN. Το σημείο λοιπόν αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό βλέπουμε ότι ε, η μέθοδος αυτή, η πολυμερής που υπάρχει και η διεθνής εκπροσώπηση έχει ε, εν μέρη τουλάχιστον ε, λάβει χώρα και βλέπουμε ότι το όραμα, ή αν θέλετε το αμερικανικό όραμα το οποίο βλέπουμε για την διαφάνεια και για την πολυμερή εταιρική σχέση υφίσταται και αυτό, αυτό που, μου, που μένει ουσιαστικά να δούμε είναι πώς θα διεξαχθεί η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και της ICAN. Έχει ήδη βέβαια τοποθετηθεί και η ICAN και η Αμερικανική κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό. Πρέπει να δούμε βέβαια αν η συνεργασία αυτή μακροπρόθεσμα θα είναι βιώσιμη. Πρώτο ερώτημα όμως τώρα. Ως Ευρωπαίοι, ποιο στόχο θα πρέπει να υπερασπιστούμε κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου κατά την συνάντηση που θα γίνει με την ICAN στις Βρυξέλλες. Τι παραπάνω μπορούμε να απαιτήσουμε προς τον κύριο Κάκλινγκς και τους υπόλοιπους συμπεριγνώμονες θέτω το ερώτημα αυτό. Και το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι ότι ε, βλέπουμε ότι ε, ο ρόλος των βουλευτών είναι όλο και πιο σημαντικός. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, η έμεση επίπτωση των οδηγιών και των εκθέσεων όλων αυτών των κειμένων που καλούμεθα να εγκρίνουμε επηρεάζει την ε, διακυβέρνηση αυτή του διαδικτύου που δεν μπορεί να είναι πλέον μια κρατική κυβερνητική διακυβέρνηση αλλά πρέπει να είναι μια διακυβέρνηση που να βασίζεται στη συμφωνία όλων των συμβαλωμένων μερών. Η μέθος λοιπόν αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και στα πλαίσια αυτά ο ρόλος των βουλευτών είναι πολύ σημαντικός. Θα ήθελα λοιπόν να μας πούν οι εμπειρογνώμονές μας πώς πιστεύουν ότι θα διαρθρωθεί η συνεργασία αυτή στο μέλλον όσον αφορά την διαδικασία διακυβέρνησης διαδικτύου. Γιατί ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής πρέπει να προετοιμάσουμε και την τοποθέτησή μας για τη συνεδρίαση του Βίλνιους. Προτού περάσουμε στη νέα περίοδο, στη νέα φάση. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη των επόμενων ετών και τι θα γίνει ουσιαστικά με το IGF. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φανίστερ Ρόι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό παρακλάδι αυτό, μια καλή δυνατότητα ώστε να εμπλακεί περισσότερο το Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε και την έκθεση Τράουτμαν στο παρελθόν. Επρόκειτο και για το θέμα της ε, διοίκησης ή διακυβέρνησης. Τώρα αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας επικεντρώνεται και πολύ καλά όχι μόνο τόσο σε προϊόντα αλλά σε πτυχές της διοίκησης, της διακυβέρνησης. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι θα κάνουμε εδώ εμείς λοιπόν. Είναι μια διαδικασία μάθησης, εκμάθησης. Πρόκειται για τις θεμελιώδεις αξίες μας στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να τις επιτύχουμε, να τις εφαρμόσουμε αυτές τις αξίες, να τις υλοποιήσουμε, χωρίς να παρεκκλίνουμε ή να βασιστούμε ιδιαίτερα σε διακυβερνητικό επίπεδο ή κυβερνητικό επίπεδο γιατί πρόκειται για την προάσπιση των δικών μας θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Είχα πάει στη Σανγκάη και είδα πώς οι Κινέζοι προβληματίζονται για αυτό το θέμα. Ποια είναι τα επιχειρήματα των Κινέζων, τελείως διαφορετική η δική τους προσέγγιση από εμάς. Αν μπορούμε να προωθήσουμε το ICAN, σίγουρα είναι κάτι που μπορούμε να χαιρετήσουμε. Και πρόκειται και για το ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε να μην περάσουν όλα αυτά στα λάθος χέρια και τα διαχειρίζονται λάθος άνθρωποι έχουμε μάθει κάποια πράγματα σε αυτή τη διαδικασία μετά την Κοπενχάγη, μετά τη Σύνοδο για τις κλιματικές αλλαγές. Είδαμε, μάθαμε τι συνέβη εκεί. Πολύ κακό για το τίποτα, μεγάλος θόρυβος ε, χωρίς αποτέλεσμα. Καλό λοιπόν να εμπλακεί το Κοινοβούλιο, πιστεύω εγώ, σε αυτές τις διαδικασίες και βλέπω μια ευκαιρία και ένα ενδιαφέρον που υπάρχει. Ενδιαφέρον για τη δουλειά μας που θέλουμε να ευοδοθεί. Τώρα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το IGF ε, για αυτό το φόρμα. Έχω και μια ερώτηση όμως. Η διακυβέρνηση στο διαδίκτυο είναι σημαντική υπόθεση και αυτό το IGF είναι πολύ σημαντική υπόθεση αυτό το φόρουμ. Ε, πρέπει όμως περισσότερο τα αναπτυσσόμενα κράτη να τα εντάξουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αν δούμε χώρες της Αφρικής, πώς μπορούμε τις αφρικανικές χώρες να τις εντάξουμε, να τις εμπλέξουμε περισσότερο. Υπάρχουν πάρα, πολλές, πολλά παράπονα και ενστάσεις. Μας λένε δεν είμαστε οικονομικά σε θέση να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Στην Τινησία το είδαμε ότι και υπάρχει και βούληση να υποστηρίξουμε αυτές τις χώρες. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει μια ειδική ξεχωριστή προσφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ενταχθούν εκείνοι που έχουν κάποιες επιφυλάξεις και να μπορέσουν και εκείνοι να συμμετάσχουν όσον αφορά το IGF, αυτό το φόρουμ. Θα υπάρξει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την πτυχή. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποια λίγα λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Θα παρακαλούσα για κάποιες ερωτήσεις να μας πείτε ποιος από τους πραγματογνώμονες θα ήθελε κάτι να πει, να τοποθετηθεί. Δεν πρέπει όλοι υποχρεωτικά να τοποθετηθούν. Κάποιες ερωτήσεις σας διατυπώθηκαν. Κάποιος μπορεί να απαντήσει απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, να δώσει κάποιες απαντήσεις. Εσείς τότε μπορείτε να παρέμβετε, παρακαλώ. Τι θα μας το πείτε. Είχε και μια συγκεκριμένη ερώτηση που τέθηκε από πλευράς ε, Επιτροπής. Παρακαλώ. Ένα λεπτό όμω παρακαλώ μόνο, εντάξει. Um, um, ναι κύριε Πρόεδρε. Τρεις ομάδες ερωτήσεων είχαμε ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με το πώς διαγράφεται το μέλλον, το εγγύς και το απότερο. Κάτι με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε είναι το ζήτημα της σύμβασης με την ΑΙΑΝΑ. Ο πρέσβης αναφέρθηκε σε αυτό. Πρόκειται για μια διμερή συμφωνία που έχει η ICAN με την Αμερικανική κυβέρνηση. και όπου προβλέπεται ότι θα διοργανώνονται οι τεχνικές, αν θέλετε, λειτουργίες που έχουν να κάνουν με τους τομείς, στην εκχώρηση ονομάτων και αριθμών. Στο παρελθόν αυτό γινόταν μονομερός από τις ΗΠΑ. Έτσι έχει κατάσταση μάλλον σήμερα. Κανείς δεν θέλει να τροποποιήσει την κατάσταση αυτή, τουλάχιστον να ταράξει τα νερά, αλλά αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό, να το συζητήσουμε με του Αμερικάνου στις ε, επικαιροποιημένες κατευθύνσεις γραμμές της Κορεπέρη που Ισπανική Προεδρία λέγεται με διπλωματικό τουλάχιστον τρόπο ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ότι λύγει σύντομα η Συμφωνία Αϊάννα και λένε ότι περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ κρατών μελών και συνεργασία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να λάβει χώρα προκειμένου να διαμορφώσουμε την συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία Αϊάννα. Με πολύ ήπιο λοιπόν τρόπο έχει αρχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολείται με το ζήτημα αυτό, το ότι δηλαδή η ΑΙΑΝΑ τυχαίνει μονομερούς διαχείρισης αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα όμως κανείς δεν θέλει να ταράξει αυτή τη στιγμή τα νερά από τη μία μέρα στην άλλη. Και η στάση η οποία ακολουθείται είναι καθαρά διπλωματική. Όσον αφορά τα επερχόμενα τώρα γεγονότα, έχουμε την συνάντηση, την διάσκεψη της ICAN στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος ενδεχομένω να παρουσιάσει και την ημερήσια διάταξη εφόσον το επιθυμείτε. Όσον αφορά τώρα την IGF. Η IGF είναι πολύ σημαντικό φόρουμ από μόνο του βέβαια, γιατί πρόκειται για ένα φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν πολλές χώρες και έχει και μία στρατηγική θέση στο μοντέλο διακυβέρνησης του διαδικτύου που ακολουθούμε. Γιατί πρόκειται για ένα φόρουμ ανοιχτό, με απόλυτη ελευθερία έκφρασης, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να εκφραστεί στην IGF, μπορεί να εκφράσει οποιοδήποτε την άποψή του. Αυτό βέβαια δεν ικανοποιεί όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου, όπως καταλαβαίνετε. Η IGF δημιουργήθηκε για περίοδο 5 ετών και κλείνει σύντομα ο πενταετής αυτός πρώτος κύκλος. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει να συνεχίσει για πέντε ακόμα χρόνια την IGF. Αυτή είναι η θέση μας τουλάχιστον. Εμείς από ευρωπαϊκής πλευράς λέμε ότι μπορεί να βελτιωθεί η IGF, να γίνει λίγο πιο ορατή, να πάει περισσότερο προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βέβαια θα πρέπει να δοθούν χρήματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει χρήματα γι' αυτό και η ICAN το έχει κάνει προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν και οι αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίω η κοινωνία των πολιτών από τις χώρες αυτές. Το σημαντικό όμως είναι η IGF να συνεχίσει ως έχει, δηλαδή να είναι μία αυτορυθμιζόμενη οργάνωση, ένα αυτορυθμιζόμενο φόρουμ στο οποίο να συμμετέχουν όσο να τον περισσότερες χώρες. Δεν θα πρέπει να μπει στη γραφειοκρατία, στις γραφειοκρατικές εγκυλωτικές δομές των ΗΠΑ γιατί θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα χάσει το μοναδικό της χαρακτήρα. Πραγματικά λοιπόν η IGF κατέχει πρωταρχική θέση, πολύ σημαντική θέση στο δικό μας μοντέλο διακυβέρνησης του διαδικτύου παρακολουθούμε εκ του σύνεγγι τα όσα γίνονται εκεί και τα όσα γίνονται βέβαια και στην Γενέβη, τις σημαντικές αυτές συζητήσεις που θα γίνουν στην CSDA, στην ε, σημαντική αυτή επιτροπή των ε, Ηνωμένων Εθνών που θα συνεδριάσει σε δύο εβδομάδες. Βρισκόμαστε πάντως σε μια κρίσιμη αυτή τη στιγμή φάση για το μέλλον της IGF. Παρακολουθούμε όμως την κατάσταση, είμαστε έτοιμοι, γνωρίζουμε ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Κύριος Πρέσβης, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω για το θέμα της IGF, εφόσον ο εκπρόσωπος της Επιτροπής το κάλυψε. Απλώς μια παρατήρηση για τη δήλωση της κυρίας Τροτμάν. Είναι μια απίστευτη εξέλιξη αυτή που είχαμε τα τελευταία δέκα χρόνια σε επίπεδο ICAN. Όμως και στο εσωτερικό της ICAN οι επιδόσεις έχουν εξελιχθεί σε απίστευτο βαθμό. Δεν θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά τη σημασία των αναθεωρήσεων. Είναι σημαντικές γιατί δείχνουν ότι η ICAN αποκτά πλέον μια οπτική γωνία που έχει πάντοτε υπόψη την παγκοσμιοποίηση. Αλλά το πλέον σημαντικό είναι τι επιδόσεις θα δώσει η ICAN υπό τη δέσμευση αυτή. Αυτό είναι το πιο ζωτικό και το πιο σημαντικό και το πιο θεμελιώδες. Θα πρέπει οι επιδόσεις να είναι στο επίπεδο των δεσμεύσεων της συμφωνίας. Οι αναθεωρήσεις έρχονται ως ε, συνέπεια ως επαλήθευση, αλλά πρέπει να τους πιέσουμε, να τους ενθαρρύνουμε, να δώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόζα Φάγνερ παρακαλώ έχει τον λόγο, συνάδελφός μας. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πιστεύω σίγουρα ότι είχαμε σήμερα το πρωί μια εξαιρετική, εξαιρετική συνεδρίαση οι προσκεκλημένοι μας μας έδωσαν ε, πάρα πολύ επικοδομητικές ε, πλούσιες πληροφορίες και νομίζω και πάρα πολύ ευχάριστες. Δεν νομίζω μπορεί κανείς να κάνει κάτι παραπάνω. Είναι πολλά τα προβλήματα που τέθηκαν. Τώρα δεν είναι η ώρα για να ξανανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε χρόνο. Σημείωσα εγώ και οι συνεργάτες μου όλα αυτά τα προβλήματα ώστε να τα δούμε στην έκθεση που θα πάρει την τελική της μορφή εντάσσοντας και αυτά, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της παρέμβασης της κυρίας Τράουτμαν, της Ευρωβουλευτού Τράουτμαν και του κυρίου Φανίστερ Ρόι, διότι κατέδειξαν σαφώς και αυτό μπόρεσαν να κάνουν <clears throat> τα προβλήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απασχολούν την Ευρώπη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να επιμείνω <clears throat> και να ολοκληρώσω με αυτό, διότι θεώρησα ήταν σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις, ότι η Ευρώπη, θέλω να πω, έχει μεγάλη σύγχυση και πολλές φορές είναι πολύ διχασμένη σε πολλά θέματα. Αυτή είναι η επίκριση που ε, γίνεται σε σχέση με το ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο. Τώρα έχουμε ευκαιρία με τη διακυβέρνηση, διαχείριση του διαδικτύου η Ευρώπη να είναι ενωμένη. Ενωμένη πέρα και πάνω από τα εθνικά συμφέροντα και να είναι ενωμένη και πέρα <clears throat> από τις εντάσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι το μήνυμα η φωνή, η ευρωπαϊκή ενιαία ενωμένη φωνή μέσα στη διεθνή συγκυρία σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Τώρα με το διαδίκτυο έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία για να αρθρώσουμε αυτή τη φωνή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για την προπαρασκευή, για τα έντυπα, τα έγγραφα και αυτή την ακρόαση. 6 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για τροπολογίες, για να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προπαρασκευή, ευχαριστώ για την ε, ε, διάσκεψη αυτή και για τους ε, προσκεκλημένους που ήρθαν και τη συμμετοχή τους. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση και θα ξανασυναντηθούμε στις 3.